Bene, colleghi. Grande Britta. Συνάδελφοι. Allora, colleghi, possiamo... Συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. κηρύσω την έναρξη της συνεδρίασης, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι έχει εγκριθεί. Σημείο 2. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Η σημερινή μας συνάντηση μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Έχουμε διερμηνία διαθέσιμη σε 19 γλώσσες. Ξεκινάμε με το σημείο 3, λοιπόν. Υγεία των ζώων η εισηγήτρια, η αντιπρόεδρος Μάριτ Πόλσον. Ξεκινάει η συζήτηση και επειδή υπήρξε ένα μεγάλο αριθμό τροπολογιών, όχι μόνο για αυτό το κείμενο, αλλά για ολόκληρη τη δέσμη για την υγεία των ζώων και των φυτών, αποφασίσαμε να εκμεταλλευτούμε τη σημερινή ευκαιρία για να συζητήσουμε όλε τι τροπολογίε. Προκειμένου να υποστηρίξουμε του εισηγητέ, του κοιόδη εισηγητέ δηλαδή, και να δούμε κατά πόσο μπορούν να εξυπηρεθούν συμβαστικέ λύσει. Με απότερο στόχο να διευκολυνθεί η ψηφοφορία που όπω ξέρετε προβλέπεται για τι 11 Φεβρουαρίου της ερχόμενης, του ερχόμενου διαστήματο. Οι τροπολογίε για την έκθεση Πόλσεν ήταν 785, αλλά παραλάβαμε και μία λεπτομερέστατη γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντο και μία ακόμη από την Επιτροπή Αλία. Καταρχά λοιπόν, προσκαλώ Αντιπρόεδρο Πόλση να μας ενημερώσει για την ε, έκθεση και για τις τροπολογίες. Ελπίζω να έχετε βάλει τα ακουστικά σας. Αναγκάζομαι να μιλήσω σου ειδικά γιατί είναι τόσο πολύπλοκο το θέμα που προτιμώ να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, αλλά μην ανησυχείτε, θα τα λέω αργά για να με καταλάβετε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές. Πράγματι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία, ήμασταν δημιουργικοί, ήμασταν αποτελεσματικοί. Από νομικής πλευράς γνωρίζετε την πολυπλοκότητα του ζητήματος. Έχουμε 287 παραγράφους αυτού αυτό το κείμενο. Και έχουμε και 180 κατά εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο λοιπόν ήταν το όλο εγχείρημα. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια το ότι έχουμε 800 περίπου τροπολογίες. Συν της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος και της Επιτροπής Αλίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη η εξέταση της έκθεσης. Οι σκιώδες συζητητές ε, και εγώ λοιπόν επιλέξαμε ως μέθοδο εργασίας τη συζήτηση επί των αρχών. Και όταν συμφωνήσαμε πάνω στις αρχές αυτές και τις αναλύσαμε διεξοδικά, μετά αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές προτάσεις για να αποκρισταλώσουμε το οριστικό κείμενο, μελετήσαμε το αρχικό κείμενο και τις προτάσεις τροπολογιών. Να ξεκινήσω με τα κεφάλαια. Πρώτα απ' όλα ο τίτλος ε, «Υγεία των ζώων». Κατάσταση της υγείας των Μα Εδώ δεν γίνεται λόγος περί υγείας. Είναι νομικό το κείμενο για την πρόληψη και την ε, καταπολέμηση των επιζωτιών, των ζωνώσεων δηλαδή που μεταδίδονται είτε μεταξύ ζώων είτε από, ζώα σε, στους ανθρώπους. Εγώ θέλω να αλλάξει ο τίτλος του κειμένου αυτού, του νομοθετήματος αυτού, ώστε να λαμβάνεται ε, υπόψη και να γίνεται κατανοητό το πραγματικό περιεχόμενο της πρότασης αυτής. Δεύτερον, υπάρχουν ατυχή ζητήματα όπως αυτό της κλωνοποίησης. Η κλωνοποίηση όπως γνωρίζετε ήταν ένα άκρο επίμαχο ε, θέμα το οποίο δέχτηκε, για το οποίο υπήρξαν επιθέσεις και από όλες τις πλευρές, δεν έχει να κάνει όμως τίποτα με τις ε, λοιμώδεις μεταδοτικές νόσους. Δεν έχει να κάνει με την κλωνοποίηση το κείμενο αυτό. Παρότι έκανε μια πρόταση για την κλωνοποίηση πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δική μας Επιτροπή, η Επιτροπή Γεωργίας, θα συζητήσει αργότερα για αυτή την πρόταση. Δεν είναι όμως το αντικείμενο αυτής της πρότασης, παραλαμβάνω. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μεταφορά των ζώων, είναι σαφές ότι η μεταφορά των ζώων διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την μετάδοση επιζώτιων. Εδώ δεν μιλάμε για το 8 η διάρκεια δηλαδή της μετακίνησης μεταφοράς του ζώου δεν είναι το ουσιώδες εδώ. Αλλά αυτό που θα ήθελα να κάνω θα ήταν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το τι γίνεται και στις διασυνοριακές μεταφορές και στις εθνικές μεταφορές, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ουσιαστικά η διάρκεια της μεταφοράς. Η μετάδοση δεν έχει να κάνει με τα εθνικά σύνορα, ούτε με τη διάρκεια της μεταφοράς, αλλά με την ίδια τη μεταφορά. Οι ενδοκινοτικές μεταφορές πρέπει να αναφέρονται, όπως και οι μεταφορές, αλλά χωρίς να συζητούμε συγκεκριμένα περί διάρκειας. Επίσης μιλάμε για ένταση παραγωγής. Ε, εμείς θα προτιμούσαμε να γίνεται λόγος κυρίως για πυκνότητα παραγωγής τι θα πει όμως πυκνότητα παραγωγής. Είναι κάτι σημαντικό για την μετάδοση νόσων. Επίσης, έχουμε και την υγεία των μελισσών. Που παίζει το ρόλο της. Ξέρετε ότι πολλοί κτηνίατροι, εμπειρογνώμονες, έχουν γνώσεις ειδικέ για αυτό το θέμα, αλλά είναι λίγοι. Τι γίνεται επίσης με τους συντρόβιους οργανισμούς, τα εντρόβια ζώα. Και εδώ οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν αρμοδιότητες σε εξειδικευμένους τομείς και φορείς της υγείας. Έπειτα έχουμε και τα αδέσποτα που και αυτά είναι βέβαια φορείς ε, μεταδοτικών ε, νόσων, λύσα και άλλα και άλλες ζωνώσει μεταδίδονται από τα δέσποτα ζώα και πρέπει να βρούμε έναν ορισμό, τον κατάλληλο ορισμό για τα μη δεσποζόμενα ζώα όπως τα λέει ο κανονισμός. Είδα την πρόταση της κυρίας Γέγκλε για το άρθρο 4. Η πρόταση τροπολογίας της νομίζω ότι είναι καλή. Καλή συμβαστική πρόταση. Έπειτα άλλα θέματα. Τι κάνουμε με τα ζώα αυτά που ναι μεν δεν είναι άγρια ε, ζώα, αλλά επειδή δεν έχουν πλέον ε, έναν ιδιοκτήτη, έχουν κάπως ε, γίνει αδέσποτα, αν μπορώ να το πω έτσι, οπότε εκεί πρέπει να λάβουμε μέτρα για την υγεία αυτών των ζώων και θα πρέπει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις να προβλεφθούν και για την κατηγορία αυτών των ζώων. Τροπολογίες 5, 6 και 7. Τροπολογίες Σμιτ. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και άλλες ε, πτυχές της υγείας των ζώων που σχετίζονται με τα ζώα συντροφιά, που μπορεί και αυτά να μπορούν ε, δυνητικά να μεταφέρουν νόσους επιζωτίες. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για την μη εμπορική μεταφορά ζώνη συντροφιάς. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε να μην εξαιρέσουμε όλα τα ζώα συντροφιάς. Έπειτα. Τράπεζα δεδομένων ζώνη συντροφιάς. Τι κάνουμε με αυτή τη βάση δεδομένων, γιατί είναι σημαντικό να ελέγχουμε τα ζώα συντροφιά, αλλά πρέπει τον αριθμό τους να το περιορίσουμε. Πρώτα απ' όλα ε, θα έλεγα ότι τα σκυλιά θα έπρεπε να καταγραφούν σε μια διαβάση δεδομένων γιατί εκεί έχουμε και τη πιο μεγάλη κτηνιατρική εμπειρία. Έχω συζητήσει με κτηνιάτρους και Με ρώτησαν και αν υπάρχει έλεγχος της σεξουαλικής ζωής των γατιών. Τώρα ουσιαστικά δεν ξέρουμε να σας πω τι γίνεται ούτε με τα, με τα σκυλιά ούτε με τα γατιά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν. Πρέπει να δημιουργήσουμε βάσεις δεδομένων για να αποφύγουμε την μετάδοση ασθενειών. Υπάρχουν και άλλα επίμαχα θέματα. Μικροβιακή αντοχή, αντοχή στα αντιβιωτικά και στα μικρόβια. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Λάβαμε πάρα πολλές ε, προτάσεις τροπολογία για τα θέματα αυτά και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μας απασχολήσει η ανθεκτικότητα αυτή στα μικρόβια και στα αντιβιωτικά και τα βακτηρίδια. Η κυρία Μαγκίνες έχει καταθέσει πολλές τροπολογίες από ε, αυτού, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και τόσο σωστό να μην μιλάμε για παθογόνα, ζωοπαθογόνες ουσίες ή ε, παράγοντες. Ξέρετε, εμείς έχουμε αποκλείσει τις, ε, τα ζώα νοσοπαθογόνα και αυτό νομίζω ότι είναι μια λεπτομέρεια που μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Γι' αυτό η μικροβιακή αντοχή είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει να ελέγχουν την έγκριση των κτηνιατρικών φαρμάκων οι φορές εκμετάλλευσης για να αποφευθεί η ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Και στο άρθρο 10 ζητείται από τους φορές εκμετάλλευσης να επιδείξουν συγκράτηση, αυτοσυγκράτηση και ευφυΐα σε ό,τι αφορά τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων. Νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ και σας παρακαλώ να το σκεφτείτε, να μην ξεχνάμε αυτές τις διατάξεις Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιζωτίες και τη χρήση αντιβιωτικών στο, ε, στα ζώα, ξέρετε ότι ε, ξαπλώνει τη χρήση τους, γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη και αυτό αποτελεί έναν παράγοντα και οικονομικών προβλημάτων για τους ε, κτηνοτρόφους. Διότι υπάρχουν νόσοι που δεν έχουν καταλογραφηθεί, δεν έχουν καταγραφεί ω μεταδοτικέ, αλλά δεν πρέπει να τι ξεχνάμε παρόλα αυτά, δεν πρέπει να τι αφήνουμε εκτό. Άρα είναι σημαντικό να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν συστήματα, τέλο να έχουν στη συστήματα, τα οποία θα του επιτρέπουν να διαχειρίζονται τέτοιε νόσου, οι οποίε δημιουργούν ε, πολλά κακά σήμερα στη γεωργία και στην κτηνοτρόφια. Αυτό πάντα σε ό,τι αφορά την αντιθεκτικότητα, την αντοχή στα αντιβιωτικά. Προειδοποιούμε λοιπόν, το έχουμε κάνει και κατά το παρελθόν. Το κείμενο αυτό, επαναλαμβάνω, δεν αφορά την υγεία των ζώων. Το γνωρίζουμε. Όλοι όσοι γνωρίζουν την κατάσταση και έχουν εμπειρία από γεωργία και από κτηνοτροφία γνωρίζουν ότι υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη σχέση που είναι προφανής μεταξύ της καλής υγείας των ζώων και της ανθεκτικότητά τους απέναντι στις λοιμώδεις μεταδοτικές νόσους, τα βακτηρίδια και τα μικρόβια. Το νοσοποιητικό μας σύστημα, ξέρετε, και αυτό σε ένα βαθμό εξαρτάται από την υγεία των ζώων, γιατί υπάρχει αλυσιδωτή αντίδραση και από την ε, ανθεκτικότητα των ζώων στα μικρόβια ή τα βακτηρίδια. Νομίζω λοιπόν ότι τα φάρμακα αυτά θα πρέπει να δίδονται μόνο όταν αυτό επιβάλλεται όχι όμως ότι θα πρέπει να γίνει και περιγραφή αναλυτική και διεξοδηγή ε, ε, από το Συμβούλιο για το πότε και πού χρησιμοποιούνται αυτά τα φάρμακα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω κατεξοδότηση πράξεων. Όταν τώρα θα ψηφίσουμε για το κείμενο αυτό θα σα υπενθυμίσω το εξή. Είναι ένα πολύπλοκο. Είναι ένα πολύπλοκο κείμενο το οποίο ουσιαστικά θα έχει επιρροή στη ζωή εκατομμυρίων αγροτών και κτηνοτρόφων στην Ευρώπη. Άρα η νομοθεσία αυτή πρέπει να είναι στο δυνατόν πιο σαφής, να είναι ευανάγνωστη, εύληπτη, κατανοητή για όσους ασχολούνται με την κτηνοτροφία ή την φροντίδα ζώων εν γέννη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι παράγραφοι ε, ορισμένες φορές τόσο πολύπλοκες που δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο το τι εννοούν και πράγματι μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση. Εκατοντάδες λοιπόν παράγραφοι αλλά και, εκατοντά... και πάρα πολλά παραρτήματα που πλήττουν την οικονομία του κειμένου και που έχουν να κάνουν πιο πολύ με την εφαρμογή διατάξεων του κειμένου. Λοιπόν, ζητώ να επιδείξουμε όλοι κοινό νου, ε, να θέλησουμε το κείμενο αυτό να είναι σαφές εύληπτο. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την κυρία Πόλσον τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή καθ' αυτή. Πρώτα απ' όλα το λόγο ζήτησε η κυρία Γέγλε και μετά ο κ. Σμιτ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω εξ αρχής την κυρία Πάλουσεν, την εισηγητριά μας. Όντως στέκει. Από την έκθεση αυτή και την ε, αρχή της συνεργασίας μας ήταν πολύ καλή η συνεργασία και με την εισηγήτρια του Σκιώδης ε, και με όλες τις ομάδες. Είναι τεράστιο το πακέτο αυτό που έχουμε μπροστά μας και πρέπει να ολοκληρώσουμε και στην τελική ανάλυση θα πρέπει να πετύχουμε καλούς συμβιβασμούς. Θα ήθελα να ξεκινήσω τονίζοντα αυτό που είπε προ το τέλο ο κ. Πάουλσεν, ότι δεν πρόκειται για έκθεση για την προστασία των ζώων, το θέμα είναι η ευημερία των ζώων, γιατί αυτό ασφαλώς έχει επιπτώσει στην υγεία και στις ε, νόσους. Και άρα όλα αυτά, ναι, μπορούν να μπουν στην έκθεση, αλλά στην κατάλληλη θέση μόνο. Και σε τελική ανάλυση χρειαζόμαστε μια έκθεση η οποία θα είναι πάρα πολύ σαφή και η οποία, και η οποία δεν θα υποστηρίξει την όλη γραφειοκρατία. Σε αυτό θα επανέλθω. Το ξέρει η κυρία Πάουλσεν. Το είπαμε και στις συναντήσεις μας, κατά τις οποίες παρέστησαν και όλες οι ομάδες. Το ΕΛΚ και εγώ συμφωνούμε με πολλές από τις προσεγγίσεις της κυρίας Πάουλσεν και στον τίτλο ξεκινάμε. Και εμείς υποστηρίζουμε την αλλαγή του τίτλου, γιατί η υγεία των ζώων είναι κάπως ασαφής ε, ως όρος και θεωρούμε ότι η πρόληψη και η καταπολέμηση των ε, ζωονόσων ε, ξεκαθαρίζει την έκθεση. Η κλωνοποίηση δεν ταιριάζει εδώ. Οι μεταφορές ζώων είναι κάτι ξεχωριστό σε ό,τι αφορά το χρονικό παράθυρο. Δεν έχει, θεωρώ, χαθεί κάτι στην έκθεση αυτή. Αυτά που είπατε για τα αντιβιώτικα και για την ε, ανθεκτικότητα σε αυτά, συμφωνούμε. Αλλά να τονίσω ότι και σε αυτή την έκθεση θα θέλα να το συζητήσουμε και να βρούμε συμβαστικές λύσεις για το πώς θα, θα μπορούσαμε να θίξουμε το θέμα των εμβολιασμών. Η κυρία Πάουλσεν δικαίως και σωστά έβαλε ένα ερωτηματικό στο τι γίνεται με τα αδέσποτα ζωά και κατά πόσον έχει νόημα να μπουν και αυτά, να συμπεριληφθούν και αυτά στην έκθεση αυτή, βλέποντας πώς έχει η κατάσταση σήμερα σε ό,τι αφορά την εκτροφή των ζώων. Ξεκαθαρίζεται αρκετά εύκολα νομίζω ότι κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Αφενός έχουμε τα ζώα καλλιέργεια, ε, τα οποία εκμεταλλεύεται κανείς, ε, η εκτροφής και είναι σαφές ότι σε αυτά απευθύνεται η έκθεση αυτή σε ό,τι αφορά δηλαδή την καταπολέμηση των ζώων όσων αυτών. Και αφετέρου έχουμε και τα ε, ζώα συντροφιά, τα οποία είναι ευθύνη κάποιου συγκεκριμένου ατόμου. Ύστερα έχουμε και τα άγρια ζώα. Έχουμε κυνηγού σε όλα τα κρατημέλη που είναι υπεύθυνοι για τα άγρια αυτά ζώα. Και ύστερα έχουμε και αυτή την διάμεση κατηγορία. Τα άγρια ζώα. Από οποιαδήποτε κατηγορία ουσιαστικά. Ζώα δηλαδή, τα οποία έρχονται σε επαφή με αδέσποτα, αλλά και με δεσποζόμενα ζώα και με τον άνθρωπο και στην υγεία, ενδεχομένως να προκαλέσουν προβλήματα. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα Μία από τις μεγαλύτερες ε, δυσκολίες είναι λοιπόν η αντέσποτη σκύλη. Πώς λοιπόν να τα αποφύγουμε τα θέματα αυτά, δεν γίνεται. Στη Γερμανία οι δεσποζόμενοι σκύλοι έχουν καταχωριστεί, φορούν ε, λουριά, δεν ξέρω τι γίνεται στα κράτη-μέλη και νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορούσαμε να θίξουμε το θέμα αυτό και μετά να συζητήσουμε το ποιο έχει την ευθύνη για ποιο ζώο. Αυτός είναι ο σκοπός. Πάντα με απότερο σκοπό την προστασία των ζώων συντροφιά. Είναι διαφορετικέ οι απόψεις μας τώρα και το διαπιστώσαμε αυτό στι συζητήσει μα σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα ε, των επισκέψεων ε, σε κτηνιατρικές υπηρεσίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να βασιστούμε σε μια αξιολόγηση κινδύνου γιατί ξέρουν ε, οι κτηνίατροι ποιες επιχειρήσεις παρουσιάζουν ποια προβλήματα. Ένα άλλο βασικό θέμα. Τα εθελοντικά προγράμματα καταπολέμησης ζωονόσων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κρατη που το κάνουν αυτό να τα υποβάλουν τα προγράμματα αυτά προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεχομένως κάποιο κράτος μέλος να μην το κάνει αυτό. Εντάξει, να την ε, ενημερώνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό συμβάλλει στη διαφάνεια, αλλά κατά τα άλλα να είναι στην ευχαίρεια του κράτους μέλους το τι θα κάνει, κατά πόσον κρίνει κάτι απαραίτητο και φυσικά θα πρέπει να έχει κάθε κράτος μέλος ε, την δυνατότητα να προστατεύει την επικράτειά του. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να προκύψει αυθαίρετα. Θα πρέπει να υπάρχει επιστημονική έγκριση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν είναι δυνατόν χωρίς επαρκής λόγους ε, οι εμπορικές σχέσεις, ιδιαίτερα στην ιστορική αγορά, να αναστέλλονται. Βλέπουμε, νομίζω, ότι πολύ σημαντικό θέμα, όλη την ομάδα μου το θεωρούν αυτό, είναι η υγεία των μελισσών. Και λοιπόν θα θέλαμε να επισέλθει και αυτό το στοιχείο στην έκθεση. Δύο θα πρέπει να είναι οι κανονισμοί και στο μέλλον, θεωρώ. Αυτό δεν είναι σαφές από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει και να αντικαταστήσει 50 υφιστάμενες οδηγίες και κανονισμούς. Αυτός είναι ο απότερος στόχος. Ε, νομίζω ότι αν είναι δύο οι κανονισμοί θα είναι λίγο πιο σαφές το τι περιλαμβάνει τι. Κανονισμός για την μην εμπορική εκτροφή ζώων συντροφιά. τον Μάιο του 2013 μετά από μακρές διαπραγματεύσεις ε, ψηφίστηκε ο σχετικό κανονισμό. Η δεύτερη έκθεση είναι ο κανονισμό για την επισήμανση των ε, ε μοσχαριών και του βοήου κρέατο. Για το βόλιο κρέα και την επισήμανση έχουμε προς μία έκθεση. Η επισήμανση καταργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έπρεπε να έχει συνεχίσει να υπάρχει. Κάτι που δεν έθιξε η κυρία Πάουλσον τώρα. Το οποίο εγώ θα ήθελα να το υπογραμμίσω παρόλα αυτά. Οι Ισπανοί μα συνάδελφοι από πλευρά του ΕΛΚ και των Σοσιαλιστών Δημοκρατών υπέβαλαν ε, μια σειρά τροπολογιών ταυτόσιμων, λέξη προς λέξη. Σας παρακαλώ, για εξηγήστε μου λοιπόν τι έχει γίνει, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό για την Ισπανία και πώς θα βρούμε μια συμβιβαστική λύση, γιατί σε τελική ανάλυση είναι ένα θέμα συμβιβασμού και πάντα είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν οι ανάγκες ενός μόνο κράτους μέλους σε θέματα τέτοιων συμβιβασμών. Και κατά δεύτερον, οι Ισπανοί από πλευρά των σοσιαλιστών υπέβαλαν και άλλη μια σειρά τροπολογίες και οι Ιταλικές τροπολογίες περιλαμβάνονται. Θα παρακαλούσα τους εισηγητές των ε, τροπολογιών ε, να ρίξουν μια ματιά προσπαθώντας να πετύχουμε μια ε, συμβαστική λύση. Αυτό με απασχολεί ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και σας κυρία Πάουλσεν. Ευχαριστούμε κύριο Σμιτ και μετά ο κύριος Καπόλας. Ευχαριστώ, Πάουλο. Θέλω και εγώ να συγχαρώ την κυρία Πόλσεν για τον τρόπο με τον οποίο εκείνη και οι συνεργάτε τη χειρίστηκαν αυτό τόσο περίπλοκο θέμα. Πάντοτε μιλάμε για καλή συνεργασία, αλλά εδώ ήταν όντω άριστη. Τα έχουμε πάει καλά ω τώρα και ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Απλώ το μέγεθο του θέματο που αυτή τη στιγμή συζητούμε έχει να κάνει με 40 κανονισμού και οδηγίε και 400, 400 νομοθεσίματα δευτερογενού νομοθεσίας. Μιλάμε για ένα τεράστιο έργο ε, ενοποίησης και της ε, νομοθεσίας. Μιλάμε για μεταδοτικές ασθένειες και ευτυχώς οι περισσότεροι συνάδελφοι προσπάθησαν να επικεντρωθούν σε θέματα που θα είχαν και κάποια προστιθέμενη αξία και παρέμεναν στην ουσία του θέματος. Για το άρθρο 1, αντιμικροβιολογική αντίσταση, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα κριτήρια για τον καταλαγοποίηση των ασθενειών στο άρθρο 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 46, πολύ καλή μεθοδολογία. Μια έκκληση για κάποιες από τις δικές μας τροπολογίες, παρακαλώ. Θέλουμε συνεργασία με τους συναδέλφους και στήριξη για τα άρθρα 1 4 για τις μελλοντικέ αποφάσεις αναθεώρησης των αποφάσεων για τον αντοπισμό των ζώων. Αυτό θα πρέπει να γίνεται με διαδικασία συναπόφασης, δηλαδή με την γνώμη του Κοινοβουλίου να εκφράζεται. Γιατί σε τριτογενή νομοθεσία δεν θα έχουμε αρκετή ε, εποπτεία και έλεγχο. Αλλά τεράστιο αντίκτυπο στους γεωργού και κτηνοτρόφους. Η, η τροπολογία μας 616 το θέμα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των προβάτων. Θα πρέπει η εκμετάλλευση γέννησης να είναι γνωστή και εκεί να υπάρχει ταυτοποίηση και μετά απευθείας κατεύθυνση στο σφαγείο. Είναι καλό να ξεκαθαριστεί με αυτή την ευκαιρία. Ε, τώρα, μια διαφωνία, άρθρο 140. Δεν είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να υπάρξουν πιστοποιητικά υγεία των ζώων για όλες τις κινήσεις ζώων μόνο για τα διασυνοριακά. Εάν αυτό περάσει, θα είναι τεράστιο το άχθος, στο γραφειοκρατικό για τις περισσότερες εκμεταλλεύσεις. Ιδίω και συγκεκριμένως επειδή πιστεύουμε ότι αυτό αφορά κυρίως θέματα της πολωνικής αγοράς. Νομίζουμε ότι με τη σωστή ότι το άρθρο αυτό θα λυνόταν καλύτερα με, το άρθρο, με καλύτερη επιβολή του άρθρου 3 του 1-2005, του κανονισμού 1-2005. Πάντως, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη γενική πορεία του κανονισμού και νομίζουμε ότι εδώ πραγματικά με αυτή τη δέσμη μέτρων έχουμε δείξει ότι μπορούμε να προσφέρουμε τη προστιθέμενη αξία για τη ζωή των πολιτών και ελπίζουμε να συνεχιστεί η καλή συνεργασία. Ευχαριστούμε, Σμιτ. Ο κύριος Καπόλας και μετά η κυρία Γιούζο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω εκ μέρους της κυρίας Μπαράτσου και προσωπικώς. Η κυρία Μπαράτσου ω ε, σχεδόν συγκέντρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών λόγω προβλημάτων με τις πτήσει δεν μπόρεσε να είναι παρούσα, αλλά μου ζήτησε να εκφράσω τη δική της άποψη αλλά και την άποψη της κυρίας Ράτσα Γκαρσία που για τον ίδιο λόγο δεν είναι παρούσα. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να πω εν παρόδο ότι η δική μας Επιτροπή πολλές φορές συμπίπτει με άλλες συνεδριάσεις όπου δεν μπορούν οι συνάδελφοι από μακρινότερες χώρες να είναι στην ώρα τους και να παρίστανται. Πάντως θέλω να εκφράσω έτσι καλλιώς τις ευχαριστίες μας στην κυρία Πόλσεν για τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε σε όλη αυτή την περίοδο με πολύ, τεχνικές, ε, πολύ τεχνικά ζητήματα που έπρεπε να εξεταστούν και έχουμε πολύ καλά θεμέλια για να βρούμε συμβαστικές λύσεις στα βασικότερα ζητήματα. Παρόλο που σε κάποια από αυτά υπάρχουν ε, διαφωνίες. Θα ήθελα να πω στην κυρία Πόλσεν ότι είναι ανάγκη η πρώτερη συμφωνία μεταξύ των ομάδων να υπάρξει ένας κατάλογος των ασθενειών, των όσων, είναι κάτι που παραμένει σταθερό. Επίσης για την κλωνοποίηση και επειδή το συζητήσαμε και θα το συζητήσουμε και στους συντονιστές ε, για την κατανομή των εισηγητών στο θέμα αυτό, δεν νομίζω ότι καλό είναι να καλυφθεί εδώ ένα θέμα τόσο περίπλοκο μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Ως προς την υγεία των ζώων χρειάζεται να βρεθεί μια συμβαστική λύση, διότι μάλλον για την ε, ευζοία των ζώων. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε για την υγεία, όχι για την ευζοία. Αλλά όπως σωστά είπε και η συγγήτρια, δεν θα πρέπει να προκαλέσουμε σύγχυση μεταξύ των δύο θεμάτων. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα εθελοντικής εκρίζωσης. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει απλώς να ενημερώνουν την Επιτροπή, όχι να ζητούν εξουσιοδότηση από την Επιτροπή. Μας φαίνεται παράλογο για προγράμματα εθελοντικά να ζητούν εξουσιοδότηση, εφόσον κάποιες φορές χρειάζεται και γρήγορη, πολύ σύντομη υλοποίηση. Μην προβλέψουμε μια περαιτέρω διαδικασία που είναι και αδικαιολόγητη. Ως προς την εντοπισμό των ε, ζώων συντροφιάς νομίζουμε ότι καλό είναι όλα τα ζώα να έχουν κάποια ταυτότητα, κάποια, κάποιο εντοπισμό, αλλά δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί αυτό. Για πολλούς λόγους. Θα πρέπει λοιπόν η συμβαστική μας λύση να λαμβάνει υπόψη και τη διάσταση του ρεαλισμού που απαιτείται εδώ. Χρειάζεται μια λύση που να μας επιτρέπει να επιδιώξουμε τους επιθυμητούς στόχους για το άρθρο 14 για την ενημέρωση των πολιτών. Είναι θεμελιώδης κανόνας, αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην ε, είναι αυτοκαταστροφικός ο κανόνας αυτός, γιατί πολλές φορές θα μιλούμε για νόσους Εάν η επικοινωνιακή στρατηγική δεν είναι σωστά σχεδιασμένη, σωστά προσανατολισμένη, μπορεί να προκαλέσει ζημιές χειρότερες από την έλλειψη ενημέρωσης ή τον ίδιο την όσο. Σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις έχουμε και πάλι κάποιους συνδυασμούς, ιδίως για τις εξαιρέσεις που μπορούν να αφορούν το σύστημα ε, ταυτοποίησης όπως ισχύει, ιδίως για τα εγωπρόβατα και βοηθή. Εδώ είναι πολύ σημαντική κατηγορία και πρέπει να προσέξουμε να μην δημιουργήσουμε προβλήματα. Πρόκειται για μια τεχνικότατη έκθεση, δεν θέλω να περάσω σε περισσότερε λεπτομέρειε. Απλώ από τη δική μα και όδη εισηγήτρια και την ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών υπάρχει πλήρη προθυμία να συνεχίσουμε το διάλογο για να εξεύρουμε συμβαστικέ λύσει ισόρροπε. Επίση, να μεταφέρω κάποιε ανησυχίε τη κυρία Σιράτσα Γκαρσία, γιατί όπω υπόθηκε η Ισπανική Αντιπροσωπή έχει συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία ε, τεχνικώ θεμελιώνονται πολύ καλά θα ήθελα λοιπόν να εισακουστούν οι απόψεις της, ιδίως οι τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τη συμπερίληψη στις ε, πρωτογενής τη ε, ασθενή προτεραιότητα, ώστε να υπάρχει καλύτερο εντοπισμό. Επίση, ένα σύνολο τροπολογιών, ώστε η έννοια του χώρου σταυλισμού να οριστεί καλύτερα. Μιλάμε για αυτού του χώρου όπου τα ζώα κατοικούν, ε, διαμένουν σε εκμεταλλεύσεις κτηνοτροφίας, την τροπολογία 3, 4, 30. Επίσης, οι απαιτήσει που έχουν να κάνουν με τα άρθρα 72 και 81, με την κτηνοτροφική παρακολούθηση Αυτό θα πρέπει να υπάρχει για τις σημαντικές νόσους, όχι για τις λιγότερο σημαντικές, μόνο για τις πολύ σοβαρές περιπτώσεις. Επίσης, η συνάδελφός μας Ράτσε παρουσίασε ένα σύνολο τροπολογιών για τον εντοπισμό των ύπων, των αλόγων, ένα θέμα εξαιρετικά σοβαρό. Να υπογραμμίσω εδώ στη χώρα μου, πριν από λίγες μέρες, ζούμε μια τραγωδία με ένα άλογο το οποίο προκάλεσε ένα οδικό ατύχημα με πολλούς νεκρούς. Δεν ήταν γνωστός ο ιδιοκτήτης. Το σύστημα εντοπισμού δεν είχε λειτουργήσει. Υπήρχαν θέματα γενετικού υλικού με το άλογο αυτό. Το άλογο αυτό όμως ήταν ανεξέλεγκτο και μπορούσε να προκαλέσει, όπως είδαμε, πολύ σοβαρή ζημιέ. Θα πρέπει λοιπόν με αυτό το σύστημα υγείας να προβλέψουμε κάτι ανάλογο όπως υπάρχει τώρα και για τα βοηδή τα εγωπρόβατα. Λαμβάνοντα πρόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτού του είδους των αλόγων. Και ένα άλλο ευαίσθητο θέμα είναι η μεταφορά ζώων εντός κάποιου κράτους μέλους. Ξέρουμε ποια είναι η δυσκολία να καλύψουμε το θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητε σε κάθε κράτο μέλο ξεχωριστά. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί σε κάθε κράτο μέλο η δυνατότητα να διοργανώσει τα πράγματα όπω ε, χρειάζεται. Και πάλι, κυρία Συγκέντρη, να σα ευχαριστήσω για την εξαιρετική σα δουλειά και να σα δηλώσω την προθυμία τη ομάδα μου να βρούμε τι καλύτερε δυνατέ συμφωνίε για ένα θέμα που έχει τόσο μεγάλη σημασία για του γεωργού και του πολίτε μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Λουί. Κυρία Γιούζο και μετά κύριο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 Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς θερμά την κυρία Πάουλσεν και την κυρία Γέγκλε για τις προσπάθειες που καταβάλουν ώστε να προχωρήσει αυτή η πρόταση που είναι πράγματι άκρος πολύπλοκη λόγω ακριβώς ε, των πολλών ρυθμίσεων που πρέπει να συγχωνευτούν σε μία. Όπως και η συγγήτρια έτσι και εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει στο κείμενο να συμπεριληφθεί ένας κατάλογος νόσων προτεραιότητας. Αυτό είναι θεμελιώδη σημασία. Θέλουμε επίσης να τονίσουμε ότι η νομοθεσία αυτή αφορά τις νόσους τα προβλήματα με τις ζωονόσους, τη μετακίνηση, τη μεταφορά των ζώων κτλ. Και πράγματι αληθεύει ότι υπάρχουν πολλά θέματα που ε, αλληλεπιδρούν με την υγεία των ζώων, τη μικροβιακή αντοχή, την ε, καλή υγεία των ζώων κτλ. Για όλα αυτά όμως υπάρχουν άλλα νομοθετήματα. Θεωρώ ότι δεν είναι σκόπιμο να τα μπερδέψουμε όλα αυτά. Αν έχουμε ένα νομοθέτημα για την καλή μεταχείριση των ζώων, ας βάλουμε εκεί ό,τι έχει να κάνει με την ε, καλή μεταχείριση των ζώων. Σε ό,τι αφορά τα μικρόβια και τα αντιβιωτικά. Αυτό δεν πρέπει να ρυθμιστεί στο παρόν κείμενο γιατί υπάρχουν ρυθμίσεις και υπάρχει κοινοτικό πλαίσιο εργασίας για το θέμα αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν αυτό να είναι αντικείμενο των νέων κανόνων για τα φάρμακα που θα παρουσιαστεί σύντομα. Να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια σε διαφορετικούς κανονισμούς, γιατί τελικά δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να μπερδεύουμε τα πράγματα και να χάνουμε την ουσία. Και τελικά τρελαίνονται αυτοί οι οποίοι πρέπει να διαχειριστούν τα πράγματα και να εφαρμόσουν την νομοθεσία. Δεν θέλω βέβαια με αυτό να πω ότι δεν έχει καμία σχέση η μικροβιακή αντοχή, η ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά με την υγεία των ζώων και με την ασφάλεια των τροφίμων. Έχει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι εξαγωγέ, θέλει να ρυθμίσει τις οικονομικές ε, συνθήκες και όρου ε, των κρατών σε σχέση με τρίτε χώρε η Κομισιόν. Είμαστε αντίθετοι, διότι άλλο είναι εισαγωγέ, άλλο εξαγωγέ. Κάθε χώρα πρέπει να συνάψει τη διμερή τη σύμβαση με την τρίτη χώρα προς την οποία θα εξαγάγει τα προϊόντα της. Άρα είναι θέμα επικουρικότητας και δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί εδώ. Επίσης συμπεριλάβαμε κάποιες τροπολογίες με στόχο να υπάρξει μια διαφοροποίηση μεταξύ νόσων που απαιτούν είτε υποχρεωτική είτε θελοντική δράση. Έχουμε λοιπόν. Θα πρέπει, αν το κράτος μέλο αποφασίσει να δρομολογήσει ένα πρόγραμμα εκρίζωση ή αν επίσημα ε, θεωρείται ότι είναι απαλλαγμένο από μία νόσο. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσετε. Σε ό,τι αφορά την επισήμανση και την καταγραφή, θέλουμε οι μορφότυποι να ε, ρυθμιστούν. Βέβαια, αυτό, μάλλον αυτό ζητάει Κομισιόν, αλλά αυτό συνεπάγεται πολύ μεγάλο οικονομικό άχθο για τι επιχειρήσει. Το σημαντικό δεν υπάρχουν μητρώα, είναι τι πληροφορίε περιέχουν αυτά τα μητρώα, αυτή κατάλογη. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μα. Γιατί αυτή η ενοποίηση, η ομογενοποίηση θα δημιουργήσει νέα προβλήματα. Τέλος, δεν είναι ξεκαθαρωμένα, αλλά φαίνεται η Κομισιόν να θέλει να ρυθμίζει τις ενδοκινοτικές μεταφορές. Μα και αυτό είναι θέμα επικουρικότητας, τις μεταφορές δηλαδή ε, μεταξύ κρατών μελών. Ξέρει τα, τα κράτη-μέλη ότι πρέπει να ελέγχουν την υγεία των ζώων τους και μετά υπάρχουν και άλλα θέματα που μπορούμε να τα συζητήσουμε διμέρως. Με την κυρία Γέγκλε Έχουμε μια πάρα πολύ καλή επαφή, ανταλλαγή απόψεων και με εσά κύριε Σίγητρε, φαντάζομαι γιατί είμαστε στην ίδια, στο ίδιο μικρό Απλά υπάρχουν θέματα που πράγματι επηρεάζουν, που πράγματι είναι σημαντικά, όμως άλλη θέση έχουν. Εκεί πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και όχι εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γιούζο, ο κύριος και μετά ο, ο αντιπρόεδρος Βατσακόφσκης. Ε, πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Συζητάμε μιλάμε για τα... την υγεία των ζώων, αλλά περιέχεται και ένα στοιχείο ευημερία των ζώων και αυτό λίγο με ανησυχεί. Τι θα είναι αυτό, μια πίσω πόρτα για την απαγόρευση ε, διαφορών κτηνοτροφικών ειδών. Θα ήθελα λοιπόν να με διαβεβαιώσει η κυρία Πόλσον ότι δεν έχει κάτι τέτοιο υπόψη της να πω και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλος ιδιαίτερος ότι λυπάμαι. Ότι είμαι, ε, ξέρω ότι θέλετε να καταργήσετε το ε, κόψιμο του ράμφου των ε, πουλερικών. Ξέρετε ότι ε, κανιβαλισμός θα προκύψει στα πτηνά αν απαγορευτεί αυτό η αφαίρεση του ράμφου των πτηνών. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μην γίνονται τέτοιε ε, επεμβάσεις σε ζώα. Δηλαδή, Χωρί να έχουν παρουσιαστεί προβλήματα. Δηλαδή, τι εννοεί. Πρώτα να γίνει καλυβανισμός μεταξύ των πτηνών και μετά να απαγορευτεί, να ε, επιτραπεί εκ νέου αυτή η παρέμβαση. 106 πράξεις κάθε εξουσιοδότηση έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των οποίων θα μπορούσε να το βάλει αυτό. Ελπίζω, σας παρακαλώ λοιπόν να με διαβεβαιώσετε ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός σας. Δεν προσπαθείτε από την πίσω πόρτα να απαγορεύσετε αυτή την επέμβαση για την αφαίρεση του ράμφου των ζών. Βαζεκόφσκι και μετά η κυρία Βρυτά Ρέμερς. E, Ευχαριστώ. Είναι καλό ότι μιλάμε για το θέμα των αδέσποτων ζώων στην στρατηγική αυτή. Η στήρωση των ε, αδέσποτων, όντω όλα αυτά αποτελούν ένα βήμα προς τα εμπρός. Αν και νομίζω ότι έχει οριμάσει το πλήρωμα του χρόνου για το θέμα αυτό, τουλάχιστον σε κάποια από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερως. Προσφάτως, όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, ε, λάβαμε δραματικά email από τη Ρουμανία, από την Βοσνία Ζεγοβίνη. Η Βοσνία Ζεγοβίνη δεν είναι, στο, δεν είναι στην Ένωση, ενώ η Ρουμανία είναι μέλος της Ένωσης. Και από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει θέμα στη χώρα αυτή σε ό,τι αφορά χιλιάδες, ε, εκατοντάδες χιλιάδες ε, αδέσποτα ζώα. Βάσει των όσων έχω βρει ως τώρα, μιλάμε για μη τήρηση βασικών προτύπων για τα ζώα. Μιλάμε για την μη αξιοπρεπή αντιμετώπιση των ζώων. Είναι ένα πρόβλημα αυτό πραγματικά και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτεί κάποια ελάχιστα πρότυπα, κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές από τα κρατημέλη σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση των ζώων μεταξύ άλλων ασφαλώς και των αδέσποτων ζώων. Σήμερα αυτό επαφίεται σε κάθε κράτος μέλος. Μπορεί κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει ό,τι θέλει. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι η αξία πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στην ικανότητα να θέτει το σωστό παράδειγμα. Τουλάχιστον αυτό ίσχυε στο παρελθόν. Η αξιοπρεπής μεταχειρίση των ζώων. Και εδώ σήμερα έχουμε ένα αρνητικό παράδειγμα σε ένα από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά λοιπόν την μεταχείριση των αδέσποτων. Σημαντικό πρόβλημα. Να μην το παίρνουμε ελαφριά. Εγώ θα επισκεφθώ ο ίδιος στην ε, Ρουμανία, αύριο μάλιστα. Φεύγω και θα εξετάσω η διεισόμαση την κατάσταση και στα καταφύγια των ζώων. Καταλαβαίνω πάντως από τα στοιχεία που έχω λάβει ότι η κατάσταση είναι προβληματική και δύσκολη και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να το παραβλέπουμε αυτό και να το αντιμετωπίζουμε ελαφριά. Πρόκειται για ένα δράμα το οποίο ζουν διάφοροι ε, πλήττει πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο τα ζώα. Ήμουν στη Ρουμανία στις αρχές του Δεκεμβρίου και ξέρω ότι πολλοί φροντίζουν τα δέσποτα αυτά. Έχουν όλη την καλή θέληση, τα ταΐζουν, τα βοηθούν. Και πραγματικά κάποια από αυτά τα δέσποτα χαίρουν πολύ καλή υγεία. Αυτό αποδεικνύει το πόσο καλά τα φροντίζουν τα άτομα αυτά και τα άτομα λοιπόν αυτά δεν μπορούν παρά να μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα και να βλέπουν πώς την χάνουν μια ξεπρεπούς μεταχείριση στα ζώα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν, πιστεύω, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, να υπάρχει κάποια πρότυπα σε ό,τι αφορά τα δέσποτα. Και πάνω απ' όλα αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπορική δραστηριότητα κατά κανέναν τρόπο, γιατί θεωρώ ότι η πηγή του προβλήματος στη Ρουμανία αλλά και σε άλλα κρατημέλη, γιατί στην Πολωνία έχουμε επίσης το πρόβλημα αυτό. Δεν τα τηλεοδεικτώ τη Ρουμανία. Ξέρω και ότι στην Πολωνία και, και στην Πολωνία τα πράγματα είναι... δεν είναι καθόλου ιδανικά. Και όταν φυσικά υπάρχει χρήμα, εμπλέκονται και εταιρείε οι οποίε προσπαθούν να βγάλουν κέρδο από τα Δέσπιτα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οι εταιρείε αυτέ δεν έχουν σκοπό να επιλύσουν το πρόβλημα. Κινητήριο δύναμη είναι το κέρδο. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση για το πολύ βασικό αυτό θέμα που απασχολεί και πάρα πολλού πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ και τώρα τελευταία η Μπρίτα Ρέμες και μετά θα πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την συνάδελφο Πάουλσεν, η οποία ε, κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή. Μιλάμε για 40 νομοθετικές πράξεις και άνω. Όλα αυτά για να συνενωθούν σε μία έκθεση είναι άθλος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απλοποίηση, αλλά να μην καταπνίξει το περιεχόμενο των νομοθετημάτων αυτών. Αυτό το νέο σύστημα θα προαπαιτήσει και κάποια καινούργια γραφειοκρατία, κάποια προσαρμογή από πλευρά των επιχειρήσεων. Όλα θα πρέπει να αλλάξουν. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κοιτάζοντα λοιπόν τι γίνεται, χρειαζόμαστε μία προσέγγιση ευρωπαϊκή σε ό,τι αφορά κυρίως την πρόληψη των ζωονόσων, το 2007 η Ρωσία είχε την Αφρικανική νόσο των χείρων, δεν κατάφερε να την περιορίσει και έφτασε στην Ευρώπη πλέον η νόσος αυτή. Στη Λιθουανία πρώτα κρούσματα παρουσιάστηκαν. Αυτό καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι και σε Ευρωπαϊκή Ένωση να βρούμε από κοινού. Από την άλλη, ασφαλώς θα πρέπει να υπάρχει και ευχέρεια σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί εκεί γνωρίζουμε πιο καλά τους πόρους μας, τους γεωργούς μας, τους εκτροφείς μας και σε περίπτωση κρούσματος μπορούμε να περιορίσουμε το κρούσμα αυτό πολύ γρηγορότερα και να μην προκαλέσουμε πανικό σε όλη την Ένωση ε, επιβάλλοντας ε, πανευρωπαϊκά μέτρα, δυσανάλογα. Ύστερα σε πολλές ε, εξαγωγικές διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες σε πολλές περιπτώσεις ε, είναι επιχείρημα κατά ημών αυτό, ότι είναι πολύ διαφορετικό το σύστημα ελέγχου που επικρατεί στην Ευρώπη. Για να μπλοκαριστούν δηλαδή οι εξαγωγές μας, το οποίο την έχει και οι οικονομικές επιπτώσεις. Καταδεικνύεται λοιπόν εκ νέου η σημασία του θέματος αυτού και η σημασία της επεξεργασίας του θέματος αυτού. Θα πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά, με προσοχή, δεν σημαίνει το ότι το σύστημα είναι παλιό, το ότι είναι και άχρηστο και δεν αξίζει σε τίποτα. Να κρατήσουμε τα καλά στοιχεία από το παλιό σύστημα. Είναι σημαντικό αυτό και για την εμπιστοσύνη από πλευρά των εκτροφέων και των επιχειρήσεων. Στη μεγάλη σειρά πράξεων ε, κατά ε, είναι πραγματικά τεράστιος ο αριθμός τους. Και η εμπειρία μας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή με την αγροτική μεταρρύθμιση να μην προκαλεί έκπληξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τεράστια δυσπιστία που επικρατεί από πλευρά του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τι ε, πράξει κατά εξουσιοδότηση. Δεν είναι δυνατόν να αποφασίζουμε κάτι ε, εδώ στο Κοινοβούλιο αυτό και στην, στο επόμενο Κοινοβούλιο να ξεπερνάτε ουσιαστικά το Κοινοβούλιο. Γιατί δεν έχει συμμετάσχει στην πράξη καταξουσιοδότηση και στην κατάρτισή της και στην ε, λήψη της απόφασης. Γι' αυτό λοιπόν η τοποθέτηση του πακέτου αυτό και η επεξεργασία έτσι, τελευταία στιγμή με προβληματίζει. Μήπως θα έπρεπε σκέφτομαι να το απορρίψω εξ αρχής, ευθύ εξ αρχής, γιατί θεωρώ ότι πρόκειται για μη τήρηση των δημοκρατικών αρχών. Τέτοια τελευταία στιγμή να συζητάμε τόσο μεγάλα και βασικά θέματα και νομίζω ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να μιλήσουμε ξεκάθαρα έξω από τα δόντια. Πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν καν χρόνο να το εξετάσουν αυτό προσεκτικά γιατί προαπαιτούνται και πάρα, πολλές, ε, πάρα πολλά καθήκοντα στις χώρες τους να ενημερώσουν, να, ε, να ενημερώσουν τους πολίτες στις χώρες τους. Αντιμετωπίζουν χρονική πίεση, εν πάση περιπτώσει, συνάδελφοι. Δυσπιστώ. Και φοβάμαι μην συμφωνήσουμε για υπερβολικά πολλές πράξεις κατά και δοθεί ε, έτσι λευκή επιταγή να προσέξουμε ιδιαίτερος προκειμένου να το επισημάνουμε αυτό και στους συναδέλφους της επόμενης θετίας να προσέξουν ιδιαίτερο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Μπρίτα. Και τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Ντομάτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Πόλσεν και τους κοιότητες εισηγητές για όλη τους τη δουλειά για να βελτιώσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προφανώς θα δείξω μόνο ορισμένα από τα σημεία που έχουν αναφερθεί. Θα προσπαθήσω να σταθώ σε αυτά που περισσότεροι βουλευτές ανέφεραν και που έχουν μεγαλύτερη πολιτική σημασία. Πάνω απ' όλα ο τίτλος και το πεδίο. Ο τίτλος της πρόταση είναι Animal Health όμως η πρόταση επικεντρώνεται στις ε, μεταδοτικές νόσους. Αυτό είναι σαφές. Εάν μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον τίτλο, δεν έχουμε πρόβλημα. Προφανώς ο τίτλος πρέπει να αντικατοπτρίζει το πεδίο και το σκοπό της οδηγίας. Δεν είναι η ευζοία των ζώων. Γι' αυτό τα επιχειρήματα όπως η κλωνοποίηση, είδατε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται στο γεγονός ότι η κλωνοποίηση αποτελεί κίνδυνο για την ευζοία των ζώων. Δεν αποτελεί μέρος της πρότασης που συζητούμε σήμερα η ευζοία. Η αποτομή των, ε, του ράμφους των ε, πτηνών, των πουλερικών, των big trimming, το big trimming. Δεν ε, θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θίξει το ζήτημα αυτό μέσω σε αυτή την πρόταση. Οκτώρες για τη μεταφορά των ζώων. Παρομοίως, Ελπίζω ότι είμαστε όλοι συνεννοημένοι και σαφείς. Μεταφορά ζώου από τη Φινλανδία στις Κανάριες νήσους μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία του ζώου, αλλά για την ευζοία μάλλον των ζώων, αλλά μπορεί να μην έχει καμία σχέση με μεταδοτικές νόσους η μεταφορά από την Ολλανδία στη Γερμανία μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο επικίνδυνη, με 100 χιλιόμετρα απόσταση μόνον. Για πολύ πιο σύντομε αποστάσει λοιπόν από την σκοπιά τη υγεία των ζώων μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτερη κίνδυνη. Οπότε δεν είναι θέμα διάρκεια τη μεταφορά αυτό που φύγουμε εδώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε σκοπό να διευθετήσουμε ε, όπω πρέπει και την μεταφορά των ζώων προκειμένου να υπάρξει πρόληψη ασθενειών. Εδώ άκουσα δύο-τρει διαφορετικές απόψεις από την κυρία Γέγκλε και την κυρία Αγιούζο. Είπαν δύο διαφορετικά πράγματα αρκετά διαφορετικά. Πιστεύω ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βρει την... Ε, το, έχει βρει, το, πιστεύω, το ορθό σημείο ισορροπίας σε σχέση με τις μετακινήσεις, τις μεταφορές στο εσωτερικό ενός κράτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της κάνει λόγο για κάποιες αρχές που διέπουν τη μεταφορά των ζώων και που εφαρμόζονται ακόμη και για τις μεταφορές εντός κράτους μέλους. Προφανώς δεν μπορεί να μετακινηθεί ένα ζώο από μια εκμετάλλευση, ένα αγρόκτημα που υπάρχει κρούσμα νόσου σε μια άλλη εκμετάλλευση αγρόκτημα που δεν υπάρχει αυτό το κρούσμα, ακόμη και αν αυτή η μετακίνηση έχει να κάνει με το εσωτερικό μιας χώρας. Δεν το επιτρέπει αυτό η πρόταση. Αφήνει όμως σε απαρκές περιθώριο στις αρχές κάθε κράτους μέλους να ε, διαθετήσουν καλύτερα αυτό το είδους της μετακινήσεις. Προφανώς η διευθέτηση της, κίνησης μετακίνησης και της μεταφοράς των ζώων είναι λεπτομερέστερη και επακριβέστερη όταν μιλάμε για διακρατικές μεταφορές. Ένα άλλο θέμα που εθίγει ήταν αυτό των ζώων που είναι δεσποζόμενα ή αδέσποτα. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσω το εξή. Όπω έχει διατυπωθεί η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασίζεται στην ιδέα ότι πρέπει να ελέγχονται οι ασθένειε των ζώων. Προφανώς ο έλεγχος αυτός για ζώα τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ανθρώπου είναι κάτι που είναι πιο εφικτό. Δεν μπορεί όμως να οργανωθούμε τον ίδιο τρόπο όταν μιλούμε για ζώα τα οποία δεν έχουν κάποιο δεσπότη, κάποιον κάτοχο ή κύριο. Είναι δύο μεγάλες λοιπόν κατηγορίες. Kept και wild είναι τα ζώα, δηλαδή δεσποζόμενα και αδέσποτα. Είναι τελείω διαφορετικό ο τρόπο επιβολή των μέτρων σε αυτέ τι δύο μεγάλε αδρέ κατηγορίε. Εάν ένα πρώην αδέσποτο σκυλί αποκτήσει κάτοχο, αποκτήσει ιδιοκτήτη, τι συμβαίνει. Απλώ περνάει από την κατηγορία wild, αδέσποτο, στην κατηγορία kept. Δεσποζόμενο. Πάντοτε έχοντα κατά νου το στόχο, τον έλεγχο των ασθενειών. Τώρα, εάν μιλήσουμε για το θέμα των αδέσποτων σκυλιών, stray dogs, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση ότι το θέμα αυτό είναι σοβαρότατο. Γι' αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και γι' αυτό στρέφεται τόσο πολύ σε αυτά η κοινή γνώμη και το Ευρωκοινοβούλιο. Όμως κοιτάξαμε και τις νομικές πτυχές του θέματος. Ο Επίτροπος Μπόρτ σε μια επιστολή που απέστειλε στον Ρουμάνο Υπουργό αποσαφήνισε την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκεί λέει ο Επίτροπος Μπορτ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα ελέγχου του πληθυσμού, του αριθμού των αδέσποτων σκύλων. Αυτό γιατί τα σκυλιά δεν είναι εκτρεφόμενα ζώα, οπότε υπάρχουν και όρια. Όρια τα οποία προβλέπει το άρθρο 13 της συνθήκης. Για αυτό το λόγο, μια συζήτηση για τέτοια θέματα μου φαίνεται εύστοχη μεν, χρήσιμη, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και ποια είναι τα νομικά όρια που μα επιβάλλονται. Σε κάθε περίπτωση και πέραν τη συζήτηση αυτή που μπορεί να έχει ε, άλλο ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί τη ουσία σκοπό έχει να ελέγξει τι ασθένειε τη νόση των ζώων, όχι να προστατεύσει τι ομάδε αδέσποτων σκύλων. Το Ξαναλέω, έχει πλήρη επίγνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σοβαρότητα του θέματο αυτού, αλλά είναι εκτός του πεδίου της συγκεκριμένη πρόταση. Σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση των ζώων. Είναι ένα ζήτημα που το έχει θίξει εδώ και πολλά χρόνια ο κ. Βίκας. Ο κύριος Σμιτ, τώρα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι έχει υπερβολικά πολλές κατεξουσιοδότηση αρμοδιότητες σε αυτή την περίπτωση. Πολλές εξουσίες. Εγώ να θυμίσω απλώς το εξή. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και με άλλους ε, βουλευτές ή άλλες βουλευτές. Μα ζητούσαν μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες για την ταυτοποίηση των ζώων, ιδίω για την ταυτοποίηση των ε, εγωπροβάτων. Εξηγήσαμε ότι συχνά η πρωτογενής πράξη δεν επέτρεπε επερκή ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μπορέσει να προβλέψει εξαιρέσεις. Έχουμε χρησιμοποιήσει στην περίπτωση της συζήτησης για την ταυτοποίηση των εγωπροβάτων το μέγιστο βαθμό ευελιξίας που διαθέταμε. Αλλά αυτόν μας επέτρεπε η οδηγία ή καλύτερα ο κανονισμός που ισχύει και αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποια όρια και να θέλουμε. Γι' αυτό καλό τον κύριο Σμίτ να σκεφτεί το εξή. Δεν μπορούμε να ε, κάνουμε επικίνδυνους ελιγμούς, ούτε στόχος είναι να μειωθεί η δυνατότητα ευελιξίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα υγείας των ζώων. Η μικροβιακή αντοχή για το θέμα αυτό Προφανώς δεν προσπαθούμε με την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συγκεντρώσουμε όλες τις πολυάριθμες αυτές δράσεις που έχουμε αναλάβει τόσα καιρό τώρα για να ελέγξουμε τη μικροβιακή αντοχή. Το λέω στα πλαίσια αυτής της πρότασης για την υγεία των ζώων, στη στιγμή που βλέπουμε αυτούς που το επιθυμούν να παρουσιάζουν τη μικροβιακή αντοχή ως προς την, ε, ε, τον έλεγχο και την εκρίζωση ως μια από τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όμως άλλα μέτρα και εδώ συμφωνώ με την κυρία Αγιούζο. Υπάρχουν άλλες αρμοδιότητες που δεν ε, περιλαμβάνονται στο πεδίο της πρότασης αυτής. Θα υποβάλουμε πρόταση για τα κτηνιατρικά φάρμακα εντός λίγων εβδομάδων και εκεί θα καλύπτονται. Για τις εξαγωγές, αυτό το έθιξε πάλι η κυρία Αγιούζο, εμείς στην πρότασή μας κάνουμε ένα copy-paste επί της ουσίας, με μικρές αλλαγές, στον υφιστάμενο κανονισμό για τα τρόφιμα. Δεν επινοούμε τίποτε το καινούριο, απλώς και στην υγεία των ζώων προσπαθούμε να προ, ε, επαναπροβλέψουμε όσα προβλέπει ο κανονισμός 178 το 2002. Πρόεδρε, ελπίζω ότι υπήρξα συνοπτικός, αλλά ότι κάλυψα τα βασικότερα ζητήματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Εγώ να δώσω πάλι το λόγο στην Αντιπρόεδρο Πόλσεν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην συμφωνούμε για όλες τις λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι σιγά σιγά με αργά αλλά σταθερά βήματα θα οδεύσουμε προς μια κοινή λύση. Το, τα προγράμματα εκρίζωσης είναι εθελοντικά. Άρα, να πω και ίδια τα κράτη-μέλη να καθορίσουν τι θέλουν να κάνουν. Εν συνεχεία πρέπει να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δράσεις, τις ενεργειές τους. Δεν θα πρέπει όμως να ζητήσουν εκ των προτέρων έγκριση για αυτά τα προγράμματα εκρίζωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί απλά να ζητήσει κάποιες πληροφορίες για να καταλάβει τι γίνεται στην επικράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα μη δεσποζόμενα ζώα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι πηγή ε, λοιμόξεων. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Με ποιο τρόπο όμως, τι πρέπει να κάνουμε. Ουσιαστικά αυτή είναι και η ουσία της ερώτησής μου. Γι' αυτό θεωρώ ότι το νομικό αυτό κείμενο δεν θα πρέπει να είναι άκρος διεξοδικό, συγκεκριμένο και αναλυτικό. Έτσι θα μπορούν να έχουν κάποια περιθώρια ελιγμών τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τη μικροβιακή αντοχή, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική την ιατρική ε, φροντίδα και η μεταφορά των ζώων. Θα πρέπει να αναφερθούμε στα νομικά κείμενα, στους κανονισμούς που υφίστανται ήδη, αλλά και στους μελλοντικού κανονισμούς. Οι αρχές είναι ένα, άλλο όμως είναι οι λεπτομέρειες. Την Τετάρτη θα έχουμε τη δυνατότητα με τους κοιότητες εισηγητές ε, στη συνεδρίαση που θα έχουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση και είμαι βεβαίω ότι θα καταλήξουμε σε σημαντικούς συμβιβασμούς. Γνωρίζετε βέβαια ότι συμβιβασμός σημαίνει ότι όλοι βάζουν νερό στο κρασί τους και ότι ε, δεν ε, θα πετύχουν όλοι στο 100% αυτό που επιδιώκουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την Αντιπρόεδρο Πόλσεν. Και προχωρούμε επιτελέστηκαν σημαντικά βήματα πρόοδου πάντως και να συγχαρώ και εγώ τη Μάριτ. Και τώρα, η ψηφοφορία θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου, οπότε μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4. Σημείο 4 στην ημερησία διάταξη, προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών. Εισηγητής, ο Χίνεκ Θεϊμούν. Η πρόταση για τους επιβλαβείς οργανισμούς που πλήττουν τα φυτά έχει σκοπό να βελτιώσει την κοινή αγορά. Έχουν υποβληθεί περίπου 331 τροπολογίες μεταξύ των οποίων 34 από τον ίδιο τον εισηγητή. Ε, και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, οι οποίες την περασμένη εβδομάδα ενέκριναν τις δικές τους εκθέσεις. Να δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή για να μας πει τις λεπτομέρειες της όλης συζήτησης και μετά περνάμε στη συζήτηση. Κύριε Φεϊμόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας κάνω μια ενημέρωση για το πώς έχει κατάσταση ναι, την έκθεσή μου που έχει να κάνει με την πρόταση της Κομισιόν για τα προστατευτικά μέρα ό,τι αφορά το αφητικό αναπαραγωγικό υλικό. Είναι μια έκθεση η οποία συνετάχθη τον Οκτώβριο. Έκτοτε κατατέθηκαν πολλές τροπολογίες. ...331 τροπολογίες κατατέθηκαν μόνο από τη δική μας Επιτροπή συζητήθηκε και στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Ο κύριος Αρέστερός ήταν συγκητή από πλευράς ΕΛΚΑ. Προστατευτικά μέτρα λοιπόν κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών. Την ψηφίσαμε στην την προηγούμενη εβδομάδα, την έκθεση αυτή μέχρι στιγμής. Δεν είχαμε όλες τις ε, γνωμοδοτήσεις, άρα και όχι όλες τις τροπολογίες. Ελπίζω αυτή τη βδομάδα να λάβουμε όλες τις τροπολογίες από όλες τις επιτροπές που νομοδοτούν. Ε, τώρα, η Επιτροπή ΕΝΒΗ κατέθεσε 180 τροπολογίες και 6 συμβιβαστικές. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων συντάσσει γνωμοδότηση σε σχέση με τη νομική βάση της όλης πρότασης. Συντάκτης της γνωμοδότησης Επιτροπής Νομικών Θεμάτων είναι η κυρία Εύλιν Ρέγκνερ από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Η γνωμοδότηση τη Επιτροπή Γιούρη, βέβαια, ένα πράγμα λέει ουσιαστικά, ότι δεν θα πρέπει να αναφερόμαστε στο άρθρο 191 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δηλαδή αυτή η σωστή νομική βάση. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε πολλά ακόμη για τις ε, τροπολογίες ούτε της Επιτροπής γιου ούτε της Επιτροπής Ένβη, δεν τις ε, εξετάσαμε διεξοδικά ακόμη, όμως ορισμένες εξ αυτών ενδέχεται να είναι ταυτόσιμες. Άρα ο κατάλογος ε, της ψηφοφορίας θα συνταχθεί με πολύ μεγάλη προσοχή και ελπίζω να καταφέρουμε να τον έχουμε ολοκληρώσει μέσα στη βδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο ελπίζω να λύσουμε τα θέματα, θα έχουμε μια συνεδρίαση με τους κοιόδης συζητητές και από κοινού φαντάζομαι θα μπορέσουμε να προτείνουμε συμβαστικές προτάσεις όπου αυτό είναι δυνατόν. Στην τελευταία μας συνεδρίαση ήδη εντοπίσαμε τέσσερις όμως μόνο τομείς μέσω των τροπολογιών ε, εκεί μπορούμε να βρούμε κάποιους συμβιβασμούς. Αυτά για τις, επιτρο... για τις τροπολίες Επιτροπής Άκρης. Ό,τι αφορά την Επιτροπή ΕΝΒΗ, επειδή δεν είχαμε στη διάθεσή μας τροπολογίες, δεν καταφέραμε να τις μελετήσουμε. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα να τις εξετάσουμε και να εκπονήσουμε συμβιβαστικές προτάσεις για όλες τις τροπολογίες που θα έχουμε λάβει μέχρι τότε. Θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε αποδεκτούς συμβιβασμούς, τουλάχιστον για την μεγάλη πλειοψηφία των μελών της ομάδας μας, έτσι ώστε να μειώσουμε όσο το περισσότερο το χρόνο της ψηφοφορίας. Δυστυχώς όμως δεν νομίζω ότι θα έχουμε και μεγάλο αριθμό συμβαστικών τροπολογιών. Όπως προείπα, συζητήσαμε τέσσερα θέματα, τέσσερις τομείς και νομίζω ότι δεν θα είναι δέκα, πάνω πάνω από δέκα οι συμβιβασμοί, διότι οι τροπολογίες είναι πολύ ετερόκλητες, ε, διαφορο διαφορετικές ε, η μία από την άλλη και δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο να τις συμβιβάσουμε σε πολλές περιπτώσεις. Άρα μάλλον έχουμε μπροστά μας ε, μια μακρό, μακρά ψηφοφορία. 500 τροπολογίε θα χρειαστεί να τεθούν σε ψηφοφορία. Έτσι έχουν λοιπόν τα πράγματα. Σε τεχνά την εκθεσή μου την προσεχή Τρίτη θα ήθελα να διοργανώσω μια ακόμη συνάντηση με τους συντονιστές, τους σκιώδεις εισηγητές μάλλον, για να συζητήσουμε μαζί την ακριβή διατύπωση των ε, συμβιβασμών. Αλλά και τη λίστα ψηφοφορίας. Είναι ένα θέμα η λίστα ψηφοφορία και πώς θα ομαδοποιήσουμε σε δέσμε τι τροπολογίε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης, το πιο αμφιλεγόμενο ή τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα ε, είναι πολλά, αλλά τρία είναι τα βασικά, τα βασικά προβλήματα. Είναι ε, το εδαφικό πεδίο εφαρμογή του όλου πακέτου, το κατά πόσον θα ισχύει για όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα εξαιρεθούν κάποιες περιφέρειες από το πεδίο εφαρμογή. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει την εξουσία να τροποποιεί τον αριθμό των ε, επιβλαβών οργανισμών ή θα εγγραφεί ε, στην νομοθεσία ο κατάλογος, θα συμπεριφθεί μάλλον στην νομοθεσία και σε περίπτωση τροποποίησης, η τροποποίηση αυτή θα πρέπει να γίνεται ε, στο πλαίσιο της τακτικής, της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Τρίτο πρόβλημα είναι αν θέλουμε έναν θετικό έναν αρνητικό κατάλογο επιβλάβων για τα φυτά ουσιών. Όταν ε, μιλάμε για εισαγωγή ε, φυτών στην Ένωση, τι θέλουμε, το άρθρο 40, θέλουμε να ισχύει όχι, με άλλα λόγια, θέλουμε έναν αυστηρό κατάλογο απαγορευμένων οργανισμών που δεν μπορούν να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα είχαμε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και λιγότερο διοικητικό βάρος. Άλλος ε, τρόπος, άλλη εναλλακτική βέβαια θα ήταν όλα τα εισαγόμενα φυτά να υποβάλλονται σε έλεγχο. Θα είναι αυτό κάτι πιο αποτελεσματικό, αλλά βέβαια θα συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερο διοικητικό βάρος. Και το βάρος αυτό θα το επομίζονται στα σύνορα της Ένωσης. Τέλος πάντων, θα δούμε και τις λεπτομέρειες τη συζήτηση. Προς το παρόν σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ξεκινούμε τώρα τη συζήτηση. Έχουμε αρκετού συναδέλφου που έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριο Ταραμπέλα και μετά η κυρία Γιούζο και πάλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι κάπω ιδιαίτερε οι συνθήκε αυτή τη στιγμή, διότι δύο συνάδελφοι μου ζήτησαν ε, να μιλήσω εκ μέρου του, η κυρία Ντανσίλα και ο κύριο ε, Ανδριέ. Δεν ξέρω αν κάνω καλά που ε, παίρνω το λόγο να μιλήσω, αλλά δεν ξέρω αν θα μιλήσω εκ μέρου και των δύο ή για δικό μου λογαριασμό. Λοιπόν, εκ μέρου τη τη κυρία Ντανσίλα, τις οποίε έλαβα το κείμενο πριν από μία ώρα από τη συνεδρίασή μας, θα σας τα πω αγγλικά. Ως και όδηση συγγήτρια για τους σοσιαλιστές στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα ε, το οποίο συζητούμε εδώ, καλωσορίζουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα προστατευτικά ε, μέτρα κατά των επιβλαβών οργανισμών ε, για τα φυτά. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς τους οργανισμούς που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία ή την βιομηχανία τροφίμων. Η κυρία Νταντσίλα ε, υποδεικνύει την ανάγκη να προστατεύσουμε τους ε, οικονομικούς και γεωργικούς μας σκοπούς. Τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα παράσιτα στα φυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την πρόπτικη της ε, προστασίας των σύνορων και των οικονομιών μας όμω, αντιμετωπίζοντας ε, ζυζάνια ή παράσιτα που έρχονται εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι επιβλαβείς οργανισμοί πρέπει να αντιμετωπιστούν με κατάλληλα μέτρα, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι συμμετέχοντες, να εφαρμόζουν την αρχή της πρόληψης και της εκρίζωσης παρασίτων, ε, με έναν τρόπο βιώσιμο προκειμένου να προστατεύσουν την ανθρώπινη υγεία, την ευρωπαϊκή γεωργία και το περιβάλλον. Αυτά από την κυρία Νταντσίλα. Και τώρα για τον κύριο Αντρίο που δεν μπορεί να είναι εδώ, ο οποίος ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι παρόν, αλλά θα ήθελε να μιλήσει για τα πιο εμβληματικά σημεία της σας νομοθεσίας και πρότασης, όπου η Ευρωπαϊκή Πρόταση περιέργως δεν προτείνει αλλαγές για τον έλεγχο των εισαγόμενων φυτών και φαρμάκων κατά των επιβλαβών οργανισμών. Η σημερινή στρατηγική που έχει να κάνει με τον έλεγχο των ε, φυτών, ετών έχει εγκριθεί από το 1977 και είναι ιδιαιτέρως αποσπασματική, διότι έχει έναν αντικό κατάλογο με φυτά, τα οποία όμως θα πρέπει να υπόκεινται σε επίσημο έλεγχο τα συνοριακά σημεία ε, πριν περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να εισάγονται χωρί κανέναν έλεγχο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιούν τα κράτη-μέλη δημιουργούν πολλά προβλήματα. Τόσο για τα προϊόντα που δεν είναι αντικείμενο αποχρεωτικού ελέγχου, τα οποία ούτω ή άλλω υπόκεινται σε έλεγχο, ε, του αρνητικού καταλόγου δηλαδή, και εκεί η σημερινή στρατηγική δεν λαμβάνει ε, αρκετά υπόψη το τι γίνεται με τι τρίτε χώρε, τι χώρε τη προέλευση. Όπω η Ταϊλάνδη, η Ινδία, η Δημοκρατία του Αγίου Δομινίκου, η Νότια Αφρική και το καθεξή. Υπάρχει ε, η κατάσχεση πολλών ε, προϊόντων, έχουμε κατάσχεση πολλών προϊόντων με τροπικά είδη, με γκογιάβες, με κολοκύθες, με μπαχαρικά, με μαντιόκα, ε, που δεν είναι σε καλή κατάσταση με πολλές φορές λευκές μύγες ή άλλου είδους παράσιτα τα οποία ε, είναι επικίνδυνα στην περίπτωση των οποροκυπευτικών αυτών και γενικότερα των καρπών και των φρούτων. Ε, τα παρασιτοκτόνα λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά πάνω απ' όλο έλεγχος στα σύνορα, διότι εκτός από τα εισαγόμενα είδη υπάρχουν και έλεγχοι της υπηρεσίας για τις νόσους, της κοινωτικής υπηρεσίας, ε, Πράγματα που αποδεικνύουν ότι η επικράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την ε, εισαγωγή επιβλαβών οργανισμών προέλευσης από τρίτες χώρες δεν εξασφαλίζεται αρκετός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνει επαρκώς με την πρότασή της ε, υπόψη αυτές τις, λειτουργίε, ούτε προτίθεται να αλλάξει το ισχύον σύστημα. Απλώς ζητά αναστολή εισαγωγών κάποιων προκυπευτικών ε, προέλευσης από την Ινδία που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα με 10 είδη που εισάγονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία, η Δανία, δεν μπορώ να τις αναφέρω όλες, η Αυστρία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Λιθουανία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Σλοβακία και η Ουγγαρία. Στο πλαίσιο αυτό, ο συνάδελφος Αντριέ, προτείνει μια σειρά από ώστε να υιοθετήσει μια συνολική σφαιρική στρατηγική η Ευρωπαϊκή Ένωση για προληπτικού σκοπού, προκειμένου να επανεξετάσει του φυτογενομικού κινδύνου που προκαλούν όλα αυτά τα εισαγόμενα ήδη λαμβάνοντα υπόψη τη χώρα προέλευση και καταρτίζοντα ένα θετικό κατάλογο ειδών, των οποίων η εισαγωγή θα μπορεί να επιτρέπεται. Όσα απορροκυπευτικά ή φυτά, δεν αναφε... φυτικά προϊόντα δεν αναφέρονται σε, αυτήν, σε αυτόν τον κατάλογο, προφανώς θα πρέπει να ελέγχονται. Το ίδιο και συνθήκη για... του ΠΟΕ για τον κατάλογο κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Τώρα, αυτή η στρατηγική θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή και πιο αποτελεσματική από την ισχύουσα και να εφαρμόζεται εδώ, όπως και σε άλλους εμπορικούς μας εταίρους, η Ινδία, η Βραζιλία, το Βιετνάμ, ε, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Εκεί τα φυτικά προϊόντα θα μπορούν να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και το αντίστροφο δεν ισχύει γιατί ακριβώ δεν υπάρχει αμοιβαιότητα στους ελέγχους. Εκεί η αλυσίδα παραγωγής δεν θα μπορεί να εγκριθεί αν δεν υπάρξει πρώτερη ε, αδειοδότηση από την χώρα εισαγωγής Οπότε οι έλεγχοι θα γίνονται και σε επίπεδο χώρα ε, παραγωγή. Θα υπάρχουν λιγότεροι έλεγχοι και άχθο για μα και λιγότερε ε, ακατάλληλε προσβάσει από τα έξω προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά για τη φυτική υγεία και για να προστατεύσουμε και τα ζώα και τι ε, νόσου των ζώων. Η κυρία Πόλσεν που ήταν εισηγήτρια για το θέμα αυτό, νομίζω θα μπορεί να επιβεβαιώσει ότι είναι σωστότερη η στρατηγική αυτή. Ολοκληρώνοντα λέγοντα ότι ο κύριο Αντρία υπέβαλε 10 τροπολογίε για του ελέγχου ε, των εισαγωγών, που και συμμερίζονται με την άποψή του είναι συνεκτικές μεταξύ τους. Διότι προβλέπουν, όπως το επιθυμεί ο συγητής, κάποιες προτεραιότητες με σταδιακή υλοποίηση μέσα σε μια τριετία της νέας προληπτικής στρατηγικής για τις εισαγωγές, ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν αυτή τη νέα προσέγγιση, να μάθουν καλά το περιεχόμενο εμπνεόμενα από τα άρθρα 228 και 331 του κανονισμού για την ευζοία των ζώων και προβλέποντας μέσα για να επιδιώξουν τους στόχους που αναφέρονται εκεί. Θα σταματήσω εδώ γιατί νομίζω είπα τα βασικότερα για την συλλογιστική του κυρίου Ανδρέα και που και εγώ συμμερίζομαι, οπότε δεν θα εκφραστώ προσωπικώς, καλύφθηκα ήδη από τον συνάδελφο. Ευχαριστώ. Bene, Ευχαριστούμε Μάρκ. Αγιούζο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή Βλάμα για έναν κανονισμό που είναι παράλληλος με αυτόν για την υγεία των ζώων και δεν θέλει να έχουμε νέους επιβλαβείς οργανισμούς στην Ένωση και όσους έχουμε να τους εκριζώσουμε. Είναι σαφή η συστόχη λοιπόν. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή που είναι αντίθετο ε, στην ε, εξαίρεση των ε, εξόχως απόκεντρων περιφερειών. τελικά αντί να είναι πλεονέκτημα για αυτές, είναι σαν να τις θεωρεί κανείς τριτοκοσμικές ε, χώρες. Και αυτό δεν είναι θετικό ούτε για τις ίδιες περιφέρειες αυτές, ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε θετικό είναι να μπορούν τα ε, κράτη, να μην μπορούν μάλλον να υιοθετήσουν πιο αυστηρά μέτρα. Ε, υπονομεύεται έτσι η λειτουργία του συστήματος. Πρέπει επίσης να επαγρυπνούμε και να παρακολουθούμε και το φυτικό υλικό που εισέρχεται με ταχυδρομικές επιστολές, με δέματα ή με κάποιους ε, ταξιδιώτες που μεταφέρουν κάτι στις αποσκευές τους. Και ξέρετε ότι υπήρξε και μία ένας ιός που η τριστέτσα των εσπεριδοειδών που ήρθε στην ε, Ένωση μέσα σε μια βαλίτσα ουσιαστικά στην Ισπανία και σε άλλες χώρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, το να μπορεί να νομοθετεί Κομισιόν σε ό,τι αφορά τι εξαγωγέ σε τρίτε χώρε. Ε, είμαστε αντίθετοι και επαναλαμβάνω αυτό που ακριβώ που είπα και για τον κανονισμό περί υγείας των ζώων. Πρέπει για τις εισαγωγές να υπάρχει νομοθεσία, αλλά όχι για τις εξαγωγές. Αυτό δεν μπορεί να το ρυθμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πόσο μάλλον ε, να υπάρχει αυτή των πιστοποιητικών. Σα δώσω ένα παράδειγμα. εμεί στην Ισπανία έχουμε περίπου 200 είδη μοντέλων υγειονομικών διαφορετικά, ανάλογα δηλαδή με τι διμερεί συμφωνίε που έχουμε με τι χώρε στι οποίε εξάγουμε τα προϊόντα μα. Βέβαια είμαστε σίγουρα ε, μια άκρο εξαγωγική χώρα φυτικών ε, προϊόντων. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε ναι να, να νομοθετούνται εισαγωγέ, αλλά όχι εξαγωγέ. Επίση θα θέλαμε οι επιβλαβείς, ε, τον, ε, οι επιβλαβείς οργανισμοί ε, να εισαχθούν ή το πρέπει να οδηγήσουν σε καρατίνα είτε όχι. Αλλά σε ένα βασικό κανονισμό να υπάρχουν αυτά τα, αυτοί οι κατάλογοι. Τώρα σε ό,τι αφορά τη δημιουργία προστατευμένων ζωνών για να μην έχουμε σημαντικοί περιορισμού σημαντικού στη μετακίνηση ε, των ε, επιβλαβών οργανισμών. Αυτό δεν το θέλουμε γιατί πρώτα πρέπει να οριστούν ως ε, οργανισμοί καραντίνας αυτοί οι οργανισμοί. Επίσης, ό,τι αφορά οργανισμούς που προέρχονται από εγκεκριμένες χώρες, πρέπει εδώ να τηρηθεί ο κανονισμός για την υγεία των ζώων. Τι γίνεται με τις εισαγωγές φυτικού υλικού. Το πρόβλημα είναι ότι μπαίνουν επιβλαβείς οργανισμοί Από την Αίγυπτο μπήκε μια, ένας επευλαβής ε, οργανισμός ε, στα φινικόδετρα και έχει μεταδοθεί τώρα παντού στην Ευρώπη. Τώρα για τις ε, εγκεκριμένε χώρες. Ό,τι ισχύει για την υγεία των φυτών πρέπει να ισχύσει. Εμείς έχουμε τελείως ανοιχτό ε, τον τομέα των ε, εισαγωγών, ενώ στις ίπα, ή σε άλλες χώρες ε, υπάρχουν τρομεροί έλεγχοι ε, και περιορισμοί, ιδίως για όσους θέλουν να βάλουν, να εισαγάγουν ένα φυτικό υλικό στην στις Ηνωμένες Θέλουμε επίσης να υπάρχει πολύ μεγαλύτερος έλεγχος σε περιοχές που δεν εφαρμόζουν τα δικά μας υγειονομικά πρότυπα. Λέω για τις εισαγωγές να εφαρμόζουμε αυτά τα οποία θέλουμε να γίνονται εδώ. Όμως, καλό θα ήταν να εισάγουμε μόνο από εγκεκριμένες περιοχές και κατ' εξαίρεση από άλλες χώρες. Με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όποτε αυτό γίνεται. Και έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Όλο και λιγότερα ζυζανιοκτώνα έχουμε για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις νόσους. Ε, και οι χώρες της Νότιας Ευρώπης ε, στις χώρες αυτές δημιουργούνται πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα από τον πλαπλασιασμό των εντόμων. Αν δεν είναι εγκεκριμένη η χώρα από την οποία εισάγεται κάτι, ποιος θα το ελέγξει μετά. Σας ευχαριστώ κυρία Αγιούζο και τώρα η κυρία Ρέιμερς και μετά ο κύριος Μπουβέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επί της αρχής η έκθεση κινείται προ τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό το ομολόγο. Χρειαζόμαστε απλοποίηση και εναρμόνιση του όλου κανονισμού. Και σκοπός είναι να μειώσουμε την γραφειοκρατία για τα κράτη-μέλη και τις ε, αρμόδιες αρχές. Αλλά και για τον παραγωγό. Και για τις επιχειρήσεις. Μείωση της γραφειοκρατίας δεν σημαίνει μόνο να απλοποιήσουμε τα πράγματα στη... σε επίπεδο διοίκησης θα πρέπει αυτό να μεταφερθεί και στο τέλος της αλυσίδας. Να μετακυλιστεί αυτή η μείωση της αγραφικρατίας. Εδώ έχουμε κάποιες αμφιβολίες σε ό,τι αφορά τον κανονισμό αυτό. Γιατί οι εκτροφείς, οι επιχειρήσεις, οι εμπορευόμενοι έχουν συνηθίσει σε έναν τρόπο λειτουργίας. Κατά πόσο βελτιώνονται λοιπόν τα πράγματα για αυτούς, δεν ξέρω, πρέπει να το σκεφτούμε. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τους επιβλαβείς οργανισμούς για τα φυτά, θα πρέπει να δούμε και τι μέσα επιτρέπουμε. Γιατί όσο πιο γρήγορη και ακαριέα είναι η καταπολέμηση, τόσο πιο μεγάλη είναι και η διευκόλυνση των επιχειρήσεων. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ευελιξία. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να περιοριστεί το όριο για την ειδοποίηση. Είναι πολύ χαμηλό το όριο στην παρούσα φάση. Για παράδειγμα σε απορροκυπιαστικά, σε περίπτωση που εντοπίζονται παράσιτα, προσπαθούν να καταπολεμηθούν, προσπαθούν να τα καταπολεμήσουν αυτά με κάποιον τρόπο, γιατί ακόμα και αν δεν είναι σωστό αυτό, είναι τεράστια δράστησε ο αντίκτυπος σε περίπτωση που το δηλώσουν και ύστερα ίσως να ευθύνονται και για τους συναδέλφους ε, σε συναδέλφους εκτροφής και γεωργούς. Άρα, ίσως αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως πρόβλημα. Όσο πιο χαμηλό είναι το όριο και τόσο πιο μικρό είναι ο αντίκτυπος, τόσο πιο εύκολα θα το δηλώνουν και η γεωργείς και ύστερα ο αρνητικός στατικός κατάλογος είναι σημαντικό θέμα το πώς θα διαμορφωθεί γιατί αν καταρτιστεί ένας κατάλογος των ε, μέσων που δεν θα πρέπει να εισαγάγονται να μην ξεχνάμε ότι στην αξιοποίηση των ε, φυτών έχουμε φυτόρια και ούτω καθεξής τομείς που απευθύνονται κατευθείαν στον πελάτη αν ξαφνικά λοιπόν προσθεθούν αυτά σε μια απαγορευμένη λίστα, ξέρουμε ότι θα αυξηθεί ο κίνδυνος εισαγωγής παρασίτων. Γιατί μέσω των τουριστικών οδών θα γίνει απόπειρα τέτοιων εισαγωγών. Και θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς το αντιμετωπίσουμε αυτό. Για κάθε μέτρο λοιπόν που προτείνουμε θα πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσο είναι βιώσιμο, εφικτό. Μην προκαλέσει μια νέα αλυσίδα συμπεριφορά που θα προκαλέσει τελικά μεγαλύτερη βλάβη. Επί της αρχής νομίζω ότι θα πρέπει να πετύχουμε διαφάνεια, προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις. Δεν θα μπορεί λοιπόν με ευελιξία να αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα έτσι, αύριο αλλιώ και να μην έχουν χρόνο, το χρόνο τον απαραίτητο οι επιχειρήσεις να προσαρμόζονται. Γιατί αυτό σίγουρα θα συνεπάγεται μεγαλύτερη γραφειοκρατία και επί του συνόλου θα ήθελα να πω και για την έκθεση αυτή, γιατί με προβληματίζει ο ρυθμό των πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Προηγουμένως αναφέρθηκε ότι θέλετε πιο πολλές πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Θέλετε μεγαλύτερη ευελιξία. Να πω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι δημοκρατικά εκλεγμένη όπως το Κοινοβούλιο. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να αναπτύξει μια πολιτική ανεξαρτησία και να καταχραστεί αυτή την ευελιξία για πολιτικούς στόχους και όχι μόνο για διοικητικές τεχνικές σκοπιμότητες. Σε επίπεδο διοικητικό, μάλιστα, να υπάρχει ευελιξία, να υπάρχουν ε, πράξεις κατά εξουσιοδότησης. Αλλά υπάρχουν τομείς πολιτικοί. Και εκεί θα πρέπει να προσέξουμε να μην ε, δημιουργείται ένας παράλληλος κόσμος, γιατί εκεί θα χάσουμε την αξιοπιστία μας στους πολίτες. Θα δεσπιστήσει ο πολίτης. Δεν θα πιστέψει ότι έχουμε μια σαφή διάκριση εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας η νομοθετική εξουσία, ε, λοιπόν, είναι στα χέρια του Κοινοβουλίου, ακόμα και αν έχει ε, δυνατότητα πρωτοβουλίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να προσέξουμε, λοιπόν, γιατί πιστεύω ότι υπερβολικά μεγάλος αριθμός ε, πράξεων κατά εξουσιοδότηση ανοίγει δρόμο προς πολιτικές σκοπιμότητες και αυτό δεν το δέχομαι. Ευχαριστούμε Μπρίτα. Ο κύριος Μποβέ και μετά η κυρία Μια σύντομη παρέμβαση. Το θέμα αυτό είναι άκρο σημαντικό. Όμως πρέπει να προσέξουμε τι κάνουμε με τις εισαγωγές, γιατί μπορεί να πέσουμε και έξω. Αναφέραμε μια σειρά από χώρες προηγουμένως. Ο κύριος Ταραμπέλα τις ανέφερε εκ μέρους του κύριου Αντρίου. Εκεί μπορεί να έχουμε αμφιβολίες να προσέξουμε, μην απορρίψουμε κάποια προϊόντα που θεωρηθούν, θεωρηθεί αυτό ως κίνηση ως μια μη ένας μη φραγμός. Διότι το πρόβλημα της υγείας των φυτικών προϊόντων σε μια συγκεκριμένη χώρα πολλές φορές δεν μπορεί να μεταδοθεί σε δικές μας. Εάν τα προβλήματα λοιπόν διαφέρουν θα πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλο σύστημα ελέγχου. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τα θέματα αυτά πολύ στενότερα και να είμαστε προσεκτικοί μην κατηγορηθούμε ότι επιβάλλουμε μη δεσμολογικού φραγμούς σε θέματα υγείας των φυτών. Δεύτερη παρατήρηση για το θέμα της συνοχή και της ε, καταπολέμησης κάποιων ε, επιβλαβών οργανισμών. Συζητήθηκε ένα ζήτημα ένα κείμενο για την φυτοκαλλιέργεια την περασμένη εβδομάδα. Και καταρτήσαμε ένα ολόκληρο σύστημα για την καταπολέμηση με πολύ συγκεκριμένη εράρχηση των θεραπείων, με την ε, μηχανική ε, πρώτα απ' όλα αντιμετώπιση και τελευταία λύση ήταν τα χημικά προϊόντα. Εάν το κείμενο λοιπόν για τα φυτικά προϊόντα, για την κυπουρική ε, μιλάει με, αυτά τα, με, αυτές τις προτεραιότητες, δεν μπορεί ένα κείμενο για τη γεωργία, την καλλιέργεια φυτών να μιλάει διαφορετικά. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια κατάλληλη συμβαστική λύση ώστε την επόμενη εβδομάδα για να συμβαστούν αυτές οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και μετά ο κύριος Καπόλας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά και συμφωνώ απόλυτα με την συνάδελφό μου, την κυρία Γιούσο, για τις ανησυχίες που έχει η χώρα μου σε σχέση με το έγγραφο αυτό. Όμως θα ήθελα να εστιάσω περισσότερο στην παρέμβασή μου ε, στις περιορισμούς, μάλλον στα λάθη τα οποία κάνει η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράγματα τα οποία άπτονται της επικουρικότητας ε, προσπαθεί να τα κοινοτικοποιήσει όταν μιλάμε για κόρηση αρμοδιοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παρέμβει σε αρμοδιότητα των κρατών μελών. Για να σεβαστούμε όμως την επικουρικότητα πρέπει να εντάξουμε τον κατάλογο των ε, κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται και των υποχρεώσεων. Και εκεί συμφωνούμε ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν τι αποφάσει για το σε ποιον θα εκχωρήσουν ε, το καθήκον του ελέγχου. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να υπαγορεύεται από τις Βρυξέλλες, γιατί αυτό ουσιαστικά περιορίζει την εθνική κυριαρχία για το θέμα των ελέγχων. Επίσης, όταν μιλάμε για την, τον έλεγχο των εξαγωγών ε, κάθε κράτους μέλους ε, στις τρίτες χώρες, πάλι ε, υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της Κομισιόν, γιατί όπως και η κυρία Γιούς έχουν πάνω από 200 ε, είδη συμβάσεων, συμφωνιών ε, στην Ισπανία και εφαρμογή διμερών συμφωνιών. Τώρα να γίνει αυτή η ομιγενοποίηση όπως ζητούν κάποια μέλη αυτού του κοινοβουλίου σημαίνει ότι τελικά διακινδυνεύουμε, βάζουμε σε κίνδυνο τις πολύπλοκες διαπραγματεύσεις που κάθε χώρα χώρα φέρει σε με καθεμία από τις τρίτες χώρες. Είναι λάθος. Δεν μπορούμε να αυτοπεριορίζουμε τις δυνατότητές μας να εξάγουμε σε διάφορα κράτη μόνο και μόνο για αυτό το καπρίτσιο της εναρμόνισης που δεν είναι και ρεαλιστική η, αυτή η πρόθεση, είναι ανεδαφική. Δεν ξέρω, μπορεί μετά από κάποιες δεκαετίες να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Στο μέλλον όμως, όχι τώρα. Ε, συμφωνίες με τρίτες χώρες είναι ε, πολύ δύσκολες ε, δαπανι... Ε, χρονοβόρες και δεν μπορούμε να τις βάλουμε σε κίνδυνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες περιορισμού ή τις λίστες αυτές του καταλόγου, εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχει ένας κατάλογος με τα εδάφη, από τα οποία μπορούμε να εισάγουμε και τι μπορούμε να εισάγουμε, γιατί έτσι θα εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα του συστήματος. Ευχαριστούμε, Λουίς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω ξανά εκ μέρου τη κοιόδουσης συγγετριά μα, τη κυρία Φιλιάτσα Γκαρσία, η οποία, όπω σα είπα, δεν μπορούσε σήμερα να είναι εδώ. Σα εξήγησα και γιατί. Υποβάλαμε ένα σύνολο τροπολογιών. Πολύ αριθμέ, ιδίω σε σχέση με τα άρθρα 40, 41, 42, 45, 68. Η τροπολογίε αυτέ αφορούν δύο βασικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, όσε θέλουν να συμπεριληφθεί στη βασική πράξη ο κατάλογος των επιβλαβών οργανισμών που θα πρέπει να ορίζονται και έπειτα το θέμα των εισαγωγών, όπως εδώ σχολιάστηκαν. Θεωρούμε ότι είναι πολύ ασφαλέστερο αυτή η νομοθετική πράξη να ευθυγραμμιστεί με το σύστημα που προβλέπουμε για την υγεία των ζώων και μόλι συζητήσαμε. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει και εδώ ένας θετικός κατάλογος. Έτσι νομίζουμε μόνον μπορούν να εγκρίνονται προϊόντα, φυτικά προϊόντα από εγκεκριμένε χώρες, Άνα προϊόν και άνα χώρα. Γι' αυτό το σκοπό ελπίζουμε ότι ο εισηγητής θα μπορέσει να συμπεριλάβει τις δικές μας βασικές μέρημνες στις συμβαστικές λύσεις που φυσικά ε, από τη μορφή που θα πάρουν αυτέ θα καθορίσουν και την, τον τρόπο που θα ψηφίσουμε όταν ψηφίσει η έκθεση αυτή στην Επιτροπή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Συνάδελφοι, ε, ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Στον κύριο Ποντλέ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Το πρόβλημα της υγείας των φυτών. Πρόκειται για ένα πρόβλημα ένα θέμα που κάπως είχε παραγωνιστεί επειδή μας απασχολούσε περισσότερο η υγεία των ζώων. Εδώ και περίπου 40 χρόνια. Όμως εδώ και 10 περίπου χρόνια καταλάβαμε ότι λόγω της έκτασης που έχει πάρει το παγκόσμιο εμπόριο και η παγκοσμιοποίηση οι ασθένειες φτάνουν και στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιοι από εσάς αναφέρατε το πρόβλημα των φοινικόδοντρων που είχαν πληγεί από ένα παράσιτο, το κόκκινο αυτό, την κόκκινη ασθένεια ε, που ήρθε από την Αίγυπτο, το είδαμε και σε πορτοκαλιές και σε άλλα φυτά και σε κάποιες περιπτώσεις σε ορισμένα είδη της Πορτογαλίας βλέπουμε ότι οι ασθένειες αυτές που έρχονται πολλές φορές προέρχονται από τρίτες χώρες. Όλη η δυσκολία έγκυται στο να βρούμε την ορθή στρατηγική για να τις αντιμετωπίσουμε. Ο κύριος Ταραμπέλα, εκ μέρους του κυρίου Ανδριό, η κυρία Αγιούζο και άλλοι μίλησαν για αλλαγή της στρατηγικής για να υπάρχει μια πολιτική καταλόγου εγκεκριμένων τρίτων χωρών. Όχι ένα ανοιχτό σύστημα όπως σήμερα ισχύει, το οποίο ανταποκρίνεται στις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Προστασία των Φυτών αληθεύει ότι κάποιες τρίτες χώρες έχουν ένα σύστημα πολύ πιο αυστηρό, πολύ πιο κλειστό. Και ξέρετε ότι αν πάει κανείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, αν έχει μαζί του κανένα μήλο στη βαλίτσα, μπορεί και να ε, δεχτεί ένα πολύ αυστηρό πρόστιμο στα σύνορα. Η αλλαγή στρατηγική που προτείνεται από ορισμένα κρατημέλη έχει συζητηθεί διαμακρών και στο Συμβούλιο έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Αυτό μας προσφέρει κάποια πλεονεκτήματα, διότι θα ήταν δυνατόν να σκεφτούμε ότι θα εγκριθεί η βελτίωση ελέγχου των εισαγωγών, όμως υπάρχουν και δυσκολίες με την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, διότι είναι πάρα πολλές οι τρίτες χώρες που παράγουν φυτικά προϊόντα, διότι σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου μας στέλνουν φυτικά προϊόντα, ενώ από κρέας λόγω χάρη Έχουμε περίπου 15 χώρες παραγωγούς από τις οποίες εισάγουμε. Τα είδη που εισάγονται, τα προϊόντα αυτά είναι πολυπίκυλα μεταξύ των δημοκρατών των δημητριακών, των προσκαλλιέργεια φυτών, των καλοπιστικών, των απορροκυπευτικών. Καθένα από τα είδη αυτά μπορεί να πληγεί από επιβλαβή οργανισμό που προφανώς ε, καλύπτουν μια τεράστια, ένα τεράστιο φάσμα. Είναι πολύ μακρύς λοιπόν ο κατάλογος τρίτων χωρών, αλλά και το προϊόν ανά τρίτη χώρα που μπορεί να εισάγουμε. Δηλαδή τεράστια διοργάνωση σε επίπεδο, όπως είπε ο κ. Μποβέ, σε επίπεδο αποτίμησης του κινδύνου, αξιολόγησης του κινδύνου από την ΕΦΣΑ. Σήμερα έχουμε ένα σύστημα το οποίο έχει χαρακτηριστεί μεν ανοιχτό, αλλά μας επιτρέπει να αντιδράσουμε και άμεσα είτε στο επίπεδο της πρόληψης είτε στο επίπεδο της θεραπείας όταν θεωρήσουμε ότι προκύπτει κάποιος κίνδυνος. Εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια λαμβάνουμε μέτρα για να χειριστούμε το θέμα τρίτων χωρών, ιδίως την Ταϊλάνδη ή την Ινδία. Υπάρχουν και άλλες βέβαια χώρες. Λαμβάνουμε λοιπόν μέτρα περίπτωση, για να περιορίσουμε τις εισαγωγές ή να έχουμε ενισχυμένους ελέγχους από τις χώρες αυτές ανάλογα με τις κοινοποιήσεις που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη. Άρα, αλλαγή στρατηγικής, ναι, αλλά είναι πολύ δύσκολη και ευαίσθητη μια τέτοια καμπή. Μπορεί να υπάρξει τεράστιο διοικητικό έργο που θα πρέπει να επιτελεστεί προηγουμένω και ξέρουμε όλοι ότι οι εθνικέ αρχέ των κατών μελών, οι φυτογειονομικέ αρχέ, είναι περιορισμένες αυτή τη στιγμή και διαρκώς μειώνονται διότι σε όλα τα κρατη οι κυβερνήσεις περιορίζουν το κρατικό τους προσωπικό. Ε, δεν ε, γλιτώνουν λοιπόν ούτε αυτές οι υπηρεσίες. Δεν γλιτώνουν από τις περικοπές στον προπολογισμό. Πρόκειται λοιπόν για απόφαση πολύ δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολο να το αποφασίσει κανείς έτσι απλά. Λίγα λόγια για τις ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές αληθεύει ότι ακόμη και βάση, εάν ε, βάσει τις συνθήκες αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τέλο πάντων συμπεριλαμβάνονται, ε, η παθογένεια των φυτών στις περιοχές αυτές είναι τελείως διαφορετική. Μιλάμε για περιοχές με τροπικό κλίμα πολλές φορές. Με παράσιτα, ζυζάνια, ιούς, ε, έντομα, μύκητες, ε, τελείως διαφορετικούς από την επικράτεια τη δική μας Επίρου και με τελείω διαφορετικέ θετικέ αντιμετώπιση. Εδώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση στο επίπεδο των συναδέλφων γενική διεύθυνση Άγκρη υπάρχουν ακριβώς τα προγράμματα ΠΟΖΕΙ, τα οποία επιτρέπουν τη χρηματοδότηση πράξεων φυτογενομική δράση στις χώρε αυτέ ακόμη και αν δεν υπάρχει ανάλογη ανησυχία ή κινητοποίηση στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και λίγα λόγια για, την, για τις κατεξοσοδότηση πράξεις για τον κατάλογο των επιλαβών οργανισμών, αν θα είναι ο κατάλογος θετικός ή αρνητικός. Όντως, τα σώμα θα επέρ της ευελιξίας για να μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε, αλλά κυρίως να προσθέσουμε επιβλαβείς οργανισμούς εφόσον χρειάζεται και ανάλογα με το κατά πόσο εμφανίζονται στην κοινοτική επικράτεια. Όμως, μέσω των ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων, όχι των εκτελεστικών, των κατεξουσιοδότηση πράξεων, θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν μεγάλη εξουσία. Διότι έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε αν η Επιτροπή έχει υπερβεί τις αρμοδιότητές της, τις εξουσίες που της αναλογούν, διότι τα κριτήρια για να μπορέσουν να συμπεριληφθούν οι οργανισμοί αυτοί στον κατάλογο ορίζονται από άρθρα του κειμένου, του κανονισμού. Οπότε έχετε κάθε δυνατότητα να ενισχύσετε ή να πλουστεύσετε τα κριτήρια αυτά. Νομίζουμε λοιπόν, ιδίω για τον κατάλογο των κατεξοδότηση πράξεων, δεν πιστεύουμε ότι το ότι η Επιτροπή θέλει να ασκήσει τη δημοκρατική της εξουσία μέσω αυτού του καταλόγου, πιστεύουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Μια κάποια ευελιξία υπάρχει και με ισχυρότατο έλεγχο από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που βλέπουν κατά πόσο εργαστήκαμε ικανοποιητικός ή όχι. Αυτά κύριε Πρόεδρε, αυτά ήθελα να σας πω. Σύντομα και μετά από όσα ανέφεραν και τα μέλη της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Τιφντά. Σε αυτή τη φάση να δώσω πάλι το λόγο στον κύριο Φάγιμο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση. Πρόκειται για ένα πολύ περιπλοκό θέμα. Και όσο πιο πολύ το συζητάμε, τόσο πιο πολλά προβλήματα ανακύπτουν. Νομίζω ότι θα είναι τεράστιο το έργο που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα σε ό,τι αφορά την κατάρτιση του καταλόγου ψηφοφορίας και την εξέβρεση μιας αποτεκτής λύσης, την οποία να αποδεχτεί η πλειοψηφία της Επιτροπής μας. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να πετύχω στο στόχο αυτό και όπως έχω ήδη πει. Την επόμενη Τρίτη στο Στρασβούργο στις 2 θα γίνει η συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Θα προσπαθήσουμε να καταρτήσουμε τον κατάλογο ψηφοφορία από κοινού και θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους για την βοήθειά τους. Ευχαριστούμε κύριε Φαϊμόν. Να θυμίσω ότι η ψηφοφορία και η έγκριση της έκθεσης προβλέπεται για τις 11 Φεβρουαρίου. Και τώρα δύο λεπτά προσοχή συνάδελφοι, διότι περνάμε στο σημείο 5 για τη σημερινή συνεδρίαση παραγωγή και θέση στην αγορά θετικό αναπαραγωγικού υλικού. Ένα κείμενο για το θετικό αναπαραγωγικό υλικό. Ο εισηγητής μας είναι ο Σέργιο Πάολο Φραντσέσκο Σιλβέστρης. Να θυμίσω συνάδελφοι ότι η συζήτηση για την έκθεση αυτή όπως ξέρετε ε, είναι πολύ σημαντική γιατί η διαπρόταση είναι πολύ σημαντική και ευαίσθητη. Το είδαμε με την υποβολή 1461 τροπολογιών, μεταξύ των οποίων 90 από τον ίδιο τον εισηγητή. Μεταξύ αυτών, όπως τα ξέρετε, κάποιες τροπολογίες ζητούν να απορριφθεί, να καταψηφιστεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θυμίζω ότι το θέμα ήδη αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης ε, σε ε, συνάντηση των σχεδόν εισηγητών στην προηγούμενη Ολομέλεια του Στρασβούργου. Οι σκιώδει εισηγητέ και συντονιστέ των διάφορων πολιτικών ομάδων, όπω το πληροφορηθήκατε, τοποθετήθηκαν και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ευρεία πλειοψηφία από όλε τι πολιτικέ ομάδε για να ζητήσουμε την απόρριψη της πρότασης αυτής με την προβολή συγκεκριμένων επιχειρημάτων, τα οποία ήταν εύστοχα. Θα συζητήσουμε τώρα αυτή την απόφαση μετά το όσα είπαν και οι συντονιστές. Νομίζω ότι εδώ στην Επιτροπή μπορούμε τώρα να τοποθετηθούμε με την παρουσία όλων των μελών της Επιτροπής, τέλος πάντων όσων κατάφεραν να είναι εδώ, ώστε να έχουμε και τη γνώμη τη δική σας. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του εισηγητή, του κυρίου Σέρδη Σιλβέστρης, ο οποίος δεν είναι εδώ. Δεν μπορούσε να παρευρεθεί, διότι έχει ένα πρόβλημα στην Ιταλία. Αλλά να θυμίσω, όπω και ο ίδιο είπε στη, της συνεδρία των συντονιστών όταν βρεθήκαμε στο Στρασβούργο, ότι θα ακολουθήσει την άποψη τη πλειοψηφία των ομάδων. Αυτήν ακριβώ την ε, θέση εξέφρασε. Οπότε ε, να εναπόκειται στην Επιτροπή μας ως σώμα των ε, βουλευτών να αποφασίσει. Οι συντονιστές αυτό αποφάσισαν άλλωστε να το συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή και θα το ξανασυζητήσουμε στη δική μας συναντρίαση μετά την Επιτροπή της Ολομέλης, την συνοδηγητή της Ολομέλης της Επιτροπής. Πρέπει να δούμε αν θα πάρουμε αυτή την απόφαση για λόγους που ήδη αναφέρθηκαν, πολυπλοκότητα του κειμένου, κατεξοδότηση πράξης που πολλοί θεώρησαν ακατάλληλες όταν συζητήσαμε σε επίπεδο συντονιστών Ανοίγουμε λοιπόν τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Ήδη κάποιοι έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των αγορητών και να θυμίσω ότι συζητούμε σε γενικέ γραμμέ και την απόφαση θα τη λάβουμε στην συνεδρίαση των συντονιστών. Η Μπρίτα Ρέιμερ ζήτησε το λόγο, μετά ο κύριο Μποβέ και ούτω καθεξή. Μπρίτα. Ευχαριστώ. Έχω ένα θέμα επί τη αρχέ για το κατά πόσον ε, υπάρχει νόημα να γίνει συζήτηση μετά από συζήτηση των αρμόδιων και δεν είναι καν εδώ πέρα και ο κύριος Λιβέθρης. δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα να το συζητήσουμε μήπως ε, να το αναβάλουμε να ε, συνεδριάσουν πρώτα και να βρουν μια συμφωνία οι αρμόδιοι δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε και τέλος πάντων δεν καταλαβαίνω τι υποτίθεται πρέπει να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Μπρίτα. Ε, συνάδελφοι, ευχαριστούμε Μπρίτα, αλλά στη συνεδρία των συντονιστών είχαμε προβλέψει το σημείο αυτό στην εμεσαία διάταξη τη σημερινή ακριβώ συζήτηση, διότι είναι ένα θέμα νομοθεσία πολύ σημαντικό. Όμω η απουσία του κυρίου Σιλβέστρη κάνει ακόμη πιο εύστοχη την παρέμβασή σου. Το λέω σε όλου του παρεμβαίνοντε, όσου έχουν ζητήσει να μιλήσουν, δεν θα το συζητήσουμε έτσι κι αλλιώ στη συνεδρία των συντονιστών. Εάν υπάρχουν όμω κάποιε παρεμβάσει οι οποίε θα τα απαραίτητε, δεν θα τι σταματήσω. Εσεί αποφασίζετε. Πάντω παρακαλώ τουλάχιστον τοποθετηθείτε σύντομα. Δεν είναι ανάγκη να μπούμε σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη κατά κάποιο τρόπο είναι και περιττό. Συμφωνώ, Μπρίτα. Ωστόσο, υπάρχει κατάλογος αγορητών, οπότε καλό να του ακούσουμε. Τώρα ο κύριο Μποβέ, ο κύριο Όσλεν και βλέπουμε. Euh, je pense Πράγματι είναι λίγο περίεργη η κατάσταση γιατί είμαστε μόνο 15 βουλευτές εδώ στην Επιτροπή και λείπει και ο εισηγητής. Είναι λίγο η κατάσταση λοιπόν. Βέβαια ε, πρόκειται για μια τροπολογία με πάνω από 1.300 τροπολογίες. Δεν πάμε καλά. Ε, δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Δεν μπορούμε να εργαστούμε σωστά. στην τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών υποτίθεται ότι κάτι είχε συζητηθεί και τώρα θα το ξανασυζητούσαμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η πρόταση να εξηγήσουμε ξεκάθαρα γιατί δεν μπορούμε να το συζητήσουμε όπως έχει αυτό το κείμενο στην παρούσα του δηλαδή μορφή, γιατί είναι θέμα ε, χρόνου αλλά και προφανές ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα πριν την τελευταία ολομέλεια να έχουμε ολοκληρώσει τη δουλειά μας. Όμως πιο σημαντικό είναι να περιοριστούμε στα πέντε σημεία τα οποία πρέπει να συζητηθούν στη συνεδρίες των συντονιστών, γιατί όχι και την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Και να εξηγήσουμε ξεκάθαρα γιατί ζητούμε να ψηφίσουμε είτε την απόρριψη είτε την, την παραπομπή, ανάπομπή του κειμένου αυτού. Είναι ένα θέμα τεχνικό εσωτερικό για την ψηφοφορία για το κείμενο. Υπάρχει ήδη ένα σημαντικό στοιχείο και εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω πάνω σε αυτό ποια είναι η θέση της Κομισιόν. Δηλαδή γιατί από την οδηγία περνάμε σε κανονισμό. Αυτό είναι κομβικό ερώτημα και θέμα, διότι από τη στιγμή που πηγαίνουμε από οδηγία σε κανονισμό δεν υπάρχει καμία εσωτερική δυνατότητα, δηλαδή ενώ σε επίπεδο κρατών μελών, να μπορέσουν να επεξεργαστούν αυτό το κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια επιλογή και αυτή η επιλογή δεν συζητήθηκε στο Κοινοβούλιο δεν συζητήθηκε εκ των προτέρων, αποτελεί δηλαδή μια πρόταση της Κομισιόν. Ε, τι ίσως την ε, πρόταση της αυτή Κομισιόν, ε, αλλά δεν είναι θέμα ε, απλό, είναι θέμα πολιτικής. Πώς ορίζουμε τις επιλογές μας σε θέματα σημαντικά όσο, όπως αυτό. Πώς περνάμε από την οδηγία σε κανονισμό. Αυτό έπρεπε να έχει συζητηθεί εκ των προτέρων, επί της ουσίας. Ναι, Ευχαριστώ, Ζωζέ. Μεταξύ άλλων, σήμερα έχουμε και την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε εδώ το Γενικό Διευθυντή μας, ο οποίος ε, μπορεί να μας πει και τη δική του γνώμη. Είναι ευκαιρία να έχουμε περισσότερες απαντήσεις. Συνεχίζουμε με τους εγγεγραμμένους. Αν μπορείτε σύντομα, ο κύριος Οσλίν, μετά ο κύριος Γκίλινγκ και ο κύριος Γιούζο. Σας ευχαριστώ να πω και εγώ από πλευρά της ομάδας μου ότι είναι περίεργο να κάνουμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό και να μην είναι παρόν ο εισηγητής. Ε, δεν ξέρω γιατί δεν είναι εδώ, αλλά εν πάση περίπτωση είναι σκιώδης αυτή η συζήτηση που κάνουμε. Και ουσιαστικά συμφωνούμε για μεγάλα θέματα σε ό,τι αφορά τα πράγματα που δεν μας βρίσκουν σύμφωνος για την οδηγία αυτή για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό. Θα θέλαμε να επισημάνουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θέλουμε να αλλάξει. Εντάξει, να το πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά τώρα να κάνουμε μια συζήτηση εδώ, χωρίς τον εισηγητή. Είναι παράλογο. Δεν χρειάζεται καν να ξεκινήσουμε. Μετά, στη συνέχεια, στην συζήτηση των συντονιστών μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα. Υπάρχουν και διαφορετικές νομικές απόψεις και ενδεχομένω αναπομπή. Ίσως θα μπορούσε να τοποθετηθεί επ' αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σας παρακαλώ μην κάνουμε τώρα συζήτηση με τέτοια απουσία αυτού που είναι υπεύθυνο να τα καταγράψει όλα αυτά. Ούτε οι σκιώδες συναντήθηκαν. Κλίμα αν ένας εισηγητής αναλαμβάνει μια τέτοια έκθεση, χρειάζεται μια δέσμευση, μια σοβαρότητα. Δεν το κατανοώ λοιπόν αυτό, πώς στέλνει κάποιον άλλον να μιλήσει εξ ονοματός του. Γκίρλινγκ e και μετά η κυρία Αγιούζο. Ευχαριστώ. Θα επαναλάβω αυτά που είπαν και οι υπόλοιποι. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Και δεν ξέρω καν ε, πώς βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Συζητήσαμε στο Στρασβούργο, στους Κιώδης και μας ζητήθηκε να σκεφτούμε πώς θα επιλύσουμε την κατάσταση και ο εισηγητής σε ό,τι αφορά την επίλυση της κατάστασης ούτε την προηγούμενη εβδομάδα ούτε την προηγούμενη κατάφερα να επικοινωνήσω μαζί του στις Βρυξέλλες. Ήταν αδύνατον να βρεθεί μια λύση επί της οποίας θα συμφωνούσαν οι σκιώδεις. Κανένα νόημα δεν βλέπω λοιπόν να συζητήσουμε αυτές τις τροπολογίες σε αυτή τη φάση γιατί να χάσουμε το χρόνο μας. Πρέπει πρώτα σε επίπεδο συντονιστών να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γκίρλικ και να υποφεληθούμε και αυτής τη συζήτησης. Παρ' όλα αυτά θεωρώ γιατί είναι εδώ ο γενικό διευθυντή, ο οποίο δεν παρευρέθηκε στην συνεδρία των συντονιστών. Και γι' αυτό λοιπόν γίνεται η συζήτηση αυτή και ασφαλώ θα συνεχίσει την συζήτηση. Η κυρία Γιούσο και η κυρία Καλαμπάχ στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ας ε, επωφεληθούμε τη παρουσία του Γενικού Διευθυντή για να κάνουμε κάποια σχόλια και μετά θα τον ακούσουμε. Πράγματι το πρόβλημα είναι άκρος πολύπλοκο. Δεν πρόκειται για οδηγία πλέον. Πρόκειται για 12 βέβαια οδηγίες. Να γίνει κανονισμός, να γίνουν κανονισμός και να ρυθμιστούν 11 διαφορετικοί τομείς. Να μπουν σε ένα νομιγενή κανονισμό. Άρα τα κείμενα ε, είναι κάπως ε, γενικόλογα ε, Ιδίω όμω, λαμβάνοντα υπόψη ότι πρόκειται για πολυτεχνικά θέματα. Ο κύριο Σιλβέστη ήταν μια αποκαταπληκτική έκθεση. Πρέπει να τη διαβάσουμε όλοι. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο της έκθεσης του κ. Σιλβέστρης, πολύ αμφιλεγόμενο, ορίζει τη, τα υλικά εξειδικευμένης αγοράς και λέει ε, ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αγορές, να έχουμε ένα, ε, διαφορές, δηλαδή να έχουμε ένα απλό μητρό με βάση την περιγραφή του υλικού, και ακολουθώντας τα πρότυπα των παραδοσιακών ποικιλιών για προϊόντα που παράγονται τοπικά και τίθενται στο εμπόριο σε μικρές ποσότητες με βάση το φυτικό υλικό. Το κριτήριο δηλαδή της Κομισιόν που συνδέει το υλικό ε, της εξειδικευμένης αγοράς με μικρό αριθμό επιχειρήσεων, με συγκεκριμένο κύκλο εργασιών και ε, συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων, αυτό το καταργεί αυτό το κριτήριο. Εάν βγάλουμε εκτός ε, τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις ε, που πολλούν σπόρους, στη μεγάλη τους πλειοψηφία πρόκειται για μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το 80% τουλάχιστον στη δική μου χώρα. Θα το θεωρήσουμε δηλαδή εξειδικευμένη αγορά το 80%. Καλές είναι οι προτάσεις του εισηγητή λοιπόν. Τώρα, λέει για τον κατάλογο και τα πρώτα πλήν του δασικού αναπαρικού υλικού θα πρέπει να, να ορίζονται με, όχι με κατεξοδοτική πράξη αλλά με τη συνήθεια νομοθετική διαδικασία. τι θα γίνει με το δασικό τομέα τελικά. Και υπάρχουν και πάρα πολλέ κατεξοδότητε πράξη. πάνω από 90 σε όλη την νομοθεσία. Εγώ όμω θέλω να κάνω και κάποιε άλλε παρατηρήσει για το δασικό τομέα. Ότι μπορεί να μείνει εκτό το δασικό αναπαγικό υλικό και υπάρχουν και κάποιες τρευλώσεις για τα δασικά είδη που είναι στο παράρτημα ένα που έχει να κάνει όμως μόνο ή μάλλον δεν έχει να κάνει με το δα, δασικά θέματα. Υπερβολικά πολλές είναι οι εκτελεστικές και κατ' πράξη 90%, 90% τον αριθμό συγγνώμη. Los sectores de plantas y semillas se ha del conjunto trasladándolo a una norma independiente. Υπάρχει επίσης και ένας ανεξάρτητος ε, κανόνας για τις υγειονομικές ε, πτυχές. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να το συζητηθεί, να συζητηθεί με τον κλάδο. Τώρα σε ό,τι αφορά τις ποικιλίε, είναι πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα. Ε, στα απορροκυπευτικά ήταν εθελοντικό, τώρα γίνεται υποχρεωτικό. Άρα πολύ μεγάλο άχθος για τα κράτη-μέλη. Επίσης, μεταχείριση των και εξέταση των ποικιλιών. Οι εξαιρέσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να προβλεφθούν και θα είναι και σημαντικές οι επιπτώσεις. Ούτε επίσης ορίζονται οι ποικιλίε με υποχρεωτική πιστοποίηση. Και μπορεί να ορίζονται στο μέλλον τα πράγματα με τα κατεξουσιοδότηση πράξη τη Κομισιόν αφού εγκριθεί ο κανονισμό. Και αυτό θα έχει ω αποτέλεσμα πολύ μεγάλη καθυστέρηση που θα στρεβλώσει πολλέ αγορέ και μάλιστα πολύ σοβαρά. Και επίσης αυτό που εγώ θεωρώ ίσως και το χειρότερο είναι αυτό το νέο μητρό κλώνων που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. να φτάσουμε σε κλόνους, είχαμε τα μητρώα με τις τρεις ε, υποδιαιρέσεις, αλλά να βάλουμε και τους κλόνους που χρησιμοποιούνται κάποιοι στην πράξη, σε κάποιους ε, οπορώνες ή σε κάποιους αμπελώνες. Είναι κάτι που θα περιπλέξει πολύ τα πράγματα. Μπορούμε να μην το επιβάλλουμε, πιστεύω. Και σε ό,τι αφορά τον ορισμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων, με πάνω από 10 επαλλήλους και λιγότερο από 10 εκατομμύρια τζίρο, Ουσιαστικά θα δημιουργήσουμε έτσι μια παράλληλη οικονομία, μια παράλληλη αγορά και νομίζω ότι αυτό δεν το θέλει κανείς. Αυτά, ευχαριστώ. E Ευχαριστούμε. Κάντεμπαχ και Ταραμπέλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, θα πρέπει να ομολογήσω ότι την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, την περιμέναμε με κάποια δυσπιστία, γιατί είχαμε κάποιες ε, αμφιβολίες σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία, την ελεύθερη πρόσβαση. Ε, είχαμε κάποιε ανησυχίε για τα θέματα αυτά. Μετά λοιπόν την πρώτη ανάγνωση μα δόθηκε η εντύπωση ότι ίσως με τη ρύθμιση σε επίπεδα ίσως να μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με κάποια στοιχεία. Εξετάζοντα πιο προσεκτικά την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να σας ε, ε, πω ότι το ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το θέμα αυτό και στο εσωτερικό και, στο, και εκτός κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι καταδεικνύει και ο μεγάλος αριθμός των ε, τροπολογιών 146 ότι συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλά που δεν μας βρίσκουν σύμφωνος ως βουλευτές μιλήσαμε για την επεξεργασία και την ε, ομαδοποίηση 12 οδηγίων. Αυτό που μας παρουσιάζεται εδώ είναι ένας κανονισμός. Ένας κανονισμός ο οποίος ε, σε μεγάλο βάθμο περιλαμβάνει αλλά και υπερβαίνει αυτά που περιλαμβάναν οι οδηγίες. Δηλαδή το πεδίο εφαρμογή του σημερινού κανονισμού είναι πολύ μεγαλύτερο από το πεδίο εφαρμογή των οδηγιών αρχικά. Δεν ανησυχούμε όμως μόνο σε ό,τι αφορά θέματα ε, εφαρμογής επειδή δεν υπάρχουν τόσο ε, περιθώριο σε εθνικό επίπεδο, γιατί σε επίπεδο βιοεπικοινότητας χρειάζεται διακριτική ευχαίρεια ανακράτως μέλος. Έχω λοιπόν ε, εξ ονόματος και της ομάδας μου υποβάλει μια σειρά τροπολογιών και παρόλα αυτά καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ακόμα και αν υπερψηφιστούν οι τροπολογίες αυτές που δεν έχει συμβεί ακόμα, ακόμα και αν βρούμε με τους κοιόδες συμβιβασμού, ακόμα και τότε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν πρόκειται να είναι σωστή. Είμαστε πεπισμένοι ότι δεν μπορεί να αλλάξει εκβάθρον και ότι θα πρέπει ότι δεν μπορούμε να καταλήξουμε στη σωστή αντιμετώπιση του θέματος και στη σωστή επεξεργασία του θέματος στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας σε ό,τι αφορά το πολλαπλασιαστικό υλικό. Είναι θέματα, ξέρετε, που αφορούν όλα τα φυτόρια, όλους τους καλλιεργητές, όλους όσους ασχολούνται με θέματα ε, βιοπικιλότητας και όλους όσους ε, όλους όσοι ασχολούνται με θέματα ασφάλειας τροφίμων. Προτείνω λοιπόν να αναπέμψουμε αυτή την πρόταση. Νομίζω ότι συμφωνεί και η πλειοψηφία, γιατί μόνο τότε θεωρώ ότι αυτές οι 12 οδηγίες θα μπορέσουν να ε, μετεξελιχθούν σε ένα σωστό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο. Σας καλώ λοιπόν να υποστηρίξετε αυτή την πρότασή σας. Ευχαριστώ κυρία Κάλενμπαχ, τώρα Μπέλα και μετά ο κύριος Ντέσου. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να επεκταθώ ω προ το εύστοχο του κειμένου και τι δυσκολίε του. Όμω έκθεση υπήρξε. Είχαμε μια πρόταση κανονισμού όπου θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να καλύπτονται 12 οδηγίε, πιο παλιά από το 1972, 1.400 τροπολογίε, πολλή δουλειά. Εγώ επέβαλα ο ίδιο 32 τροπολογίε σε σχέση με τις παλιές ποικιλίε, την ε, υφαρπαγή κάποιων ε, ποικιλιών, το δικαίωμα των πολύ μικρών επιχειρήσεων, αλλά πρέπει να μιλάμε και για τις μικρομεσαίες, που μπορεί να θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητε τους και να αυξήσουν και όχι να αφήσουν την αγορά των σπόρων στις πολυεθνικές. Όλα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα και έχω το εξή ερώτημα. Απόρριψη. Θα αποφασίσουν οι συντονιστές. Το θέμα είναι όμως μήπως αυτό πραγματικά ε, αποδυναμώνει τελείως την νομοθετική μας εξουσία και μάλιστα στα μάτια των πολιτών. Εάν προτείνουμε απόρριψη, τι θα κάνει η Επιτροπή. Το κείμενο που συνεχίσει να ζει και να συζητιέται στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα αλλάξει το κείμενό της. εμείς θα έχουμε χάσει την δυνατότητά μας να αλλάξουμε το κείμενο, να το βελτιώσουμε. Είναι λίγο σαν να όνειροβατούμε. Διότι η περίοδος είναι ιδιαίτερη. Θα ήθελα αυτό τον κίνδυνο να τον σκεφτούμε και να μας ενημερώσει η Επιτροπή για τις προθέσεις της. Εάν υπάρξει απόρριψη από το Κοινοβούλιο σε αυτό το στάδιο, τι θα γίνει μετά. Εγώ ανησυχώ. Θα ήθελα να μάθω τα πιθανά σενάρια. Ε, Ευχαριστώ. Μάρκ, τα είπαμε και στις συνεδρίες των συντονιστών. Αποφαθήκαμε, τοποθετηθήκαμε μάλλον. Η διαδικασία προβλέπει να εκφράσουμε γνωμοδότηση. Δεν ότι χάνουμε. Ε, έχουμε χρονική πίεση, γιατί στη δεύτερη ανάγνωση θα έχουμε λιγότερο χρόνο για να αντιδράσουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε λόγο. Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Ο κύριος Ντέις και ο κύριος Άγνιου. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ζητήσω συγγνώμη που καθυστέρησα κάπως γιατί ήθελα να ζητήσω και συγγνώμη εξ ονόματος του κυρίου Σιλβέστρης, ο οποίος για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παρευρεθεί και θα είχα ζητήσει να μην γίνει η συζήτηση αυτή σήμερα, να αναβληθεί. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες. Να τονίσω όμως αυτά που είπε η κυρία Γιούσο και η κυρία Κάλενμπαχ. Είναι όλα τόσο περίπλοκα. Ακόμα και όταν μιλάω με ενώσεις βιολογικών παραγωγών, είναι ασαφή τα πράγματα και δεν βλέπω πώς μπορούμε να τα λάβουμε όλα υπόψη εδώ όλα αυτά τα οποία προγραμματίζονται. Και αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερο ε, συνάδελφε Αγιούζο, είναι η 90 κατά εξουσιοδότηση πράξης. Μέχρι τον Απρίλιο δεν θα έχουμε συνάντηση. Μετά τον Απρίλιο δεν θα έχουμε πλέον άλλες συνεδριάσεις ε, και θα πρέπει δηλαδή να προσπιστώ τέτοιε πράξεις κατά εξουσιοδότηση, τις οποίες πολιτικώς δεν μπορώ να υποστηρίξω. Και ε, ιδιαίτερω τα θέματα που άπτονται τη χειρουργική μεταρρύθμιση ε, με ανησυχούν πολύ. Λοιπόν, με την ομάδα μου θα ζητήσουμε να τα κοιτάξουμε αυτά τα θέματα με την ησυχία μας. Είναι τόσο πολλά τα εκκρεμή ζητήματα που είπε ο συναδελφός Μποβέ είναι αναγκαίο και οι 12 οδηγίες να συμπεριληφθούν σε μία, μπορούν κάποια πράγματα να συνεχίσουν να ρυθμίζονται σε οδηγίες. Αυτό χρειάζεται πιο πολύ χρόνο. Οι σημερινές οδηγίες είναι αποδεκτές από όλους. Πολλά πολύ λίγα παραπονά. Πολλές λίγες ενστάσεις ε, έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν μία λύση, κύριε Ταραμπέλα, να ακολουθήσουμε και τη διαδικασία σωστά. Χρειαζόμαστε πληροφορίες από την νομική υπηρεσία και θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό στα πλαίσια της συνεδρίασης των συντονιστών και νομίζω ότι θα πρέπει με τη συμφωνία όλων των ομάδων να βρούμε μία λύση για την διαδικασία και μέσα στην επόμενη εβδομάδα να προτείνουμε μία σωστή λύση. E Ευχαριστούμε, Άλμπερτ. Άγνιου και μετά κλάσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επαναλάβω. Επαναλαμβάνω ότι συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Ντές. Εγώ έχω λάβει πάνω από 5.600 επιστολές για το θέμα αυτό, για το θέμα λοιπόν του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Ως τώρα κανείς δεν είχε παραπονεθεί για το θέμα αυτό. Άρα επιχειρούμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπάρχει. Όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ περιπλοκή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά υπάρχουν ε, άλλα δύο ε, στοιχεία που προκαλούν ιδιαίτερη σύγχυση και προστίθενται εδώ πέρα στη συγκεκριμένη κατάσταση, στην ε, κυβέρνηση της, του Ιωμένου Βασιλείου. Έχουμε πράσινες βίβλους, άσπρες βίβλους, το σκοτικό ο Κοινοβούλιο ενδεχομένως ε, να έχει και άλλου χρώματος ε, βίβλους, αλλά ποτέ δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοιο non-paper. Υπάρχει συζήτηση το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει συζήτηση. Μεγάλη σύγχυση προκαλείται. Δεύτερη σημείο σύγχυση. Δύο από τις τροπολογίε απορρίπτονται από τους συντριπτικού ε, βουλευτέ. Η σύγχυση από που προκαλείται η ΤΕΦΡΑ, που είναι το εκτελεστικό σκέλος της κυβέρνησης, δεν ε, συμφωνεί να απορριφθούν αυτές οι τροπολογίες. Μεγάλη σύγχυση και εδώ λοιπόν. Έχω την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πιο πολλά καθήκοντα από ό,τι μπορεί να εκτελέσει. Ό,τι είναι εντάξει, ας μην το πειράξουμε, εν πάση περιπτώσει. Κλάς και Γιάρ. Yeah, Σας ευχαριστώ, κυρία Κλάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από τη συζήτηση είναι σαφές ότι όλες οι ομάδες συμφωνούν ότι με 1.400 ε, τροπολογίες δεν μπορούμε να ε, ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα τόσο γρήγορα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να τράξω την ευκαιρία που μου δίνετε και να πω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσω και με τους συναδέλφους κάποια θέματα περιεχομένου. Να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Αγιούζο που επισήλθε σε κάποιες μεμονωμένες λεπτομέρειες, ένα άλλο θέμα, μια άλλη λεπτομέρεια να θίξω, το ετερογενές υλικό σε ό,τι αφορά την οδηγία για τη σποριά, αντιμετωπίζουμε μια σωρία νέων ορισμών και οι συνάδελφοι έχουν επιπρόσθετους ορισμούς για είδη καλλιεργιών, είδη εδάφους, όλα αυτά. Πώς θα τα εντάξουμε σε ένα σωστό πλαίσιο, σε ένα λογικό πλαίσιο στο τέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει κάποια σκέψη προς την κατεύθυνση αυτή, θα μας συνοδέψει στη διαδικασία αυτή σε ό,τι αφορά και αυτά που προτείνει για την εισαγωγή του ετερογενούς υλικού. Ως τώρα για την οδηγία για τους πόρους. Το θέμα ήταν να υπάρχουν αξιόπιστα είδη σπόρων για τους καλλιεργητές και τώρα ξαφνικά μιλάμε για μια ποικιλία διαφορετικών και διαφόρων και διαφορετικών όρων. Αυτό λοιπόν ως ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν θα μείνει και εκεί το θέμα. όλες αυτές τις τροπολογίες από κάποιον έχουν κατατεθεί. Κάτι έχει σκεφτεί αυτός που τις έχει καταθέσει. Δεν μπορούμε όλα αυτά να τα πετάξουμε στα σκουπίτια. Θα πρέπει να μπορέσουμε να εργαστούμε. Και γι' αυτό λοιπόν δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Θα πρέπει να δοθεί μια συνέχεια. Το θέμα που έδειξε και ο κύριος Ντές. Να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Κατά πόσον έχει νόημα να προσθεθούν και να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο και οι 12 οδηγίες ή μήπως να σκεφτούμε λίγο μεγαλύτερη διαφοροποίηση, απλοποίηση, απογραφειοκρατικοποίηση. Εντάξει, αλλά είναι μείωση της γραφειοκρατίας όταν οι 12 οδηγίες συνενωθούν σε μία, μήπως κάποια θέματα θα περιπλακούν περαιτέρω, γιατί δεν είναι δυνατόν να οματοποιηθούν και να μπουν σε παρατήματα από πλευράς λοιπόν βασικής δομής. Παρακαλώ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τους συναδέλφους να αναζητήσουμε μια λύση. Και σίγουρα χρειάζεται μεγαλύτερη συζήτηση από αυτή που μπορούμε να χωρέσουμε μέχρι 18 Απριλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πέτερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν μια παρατήρηση επί της αρχής. Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους οι οποίοι διατείνονται ότι αν θέλουμε να έχουμε μια σοβαρότητα ως κοινοβούλιο και αν θέλουμε να λάβουμε υπόψη και των πράξεων καταξουσιοδότησης ε, δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές μέσα στη θετία. Δεύτερο, προς θα πρέπει να βρούμε παρόλα αυτά ένα τρόπο να ανταλλάξουμε απόψεις Για να μην ξεκινήσουν από το μηδέν τελικά οι συνάδελφοι επόμενη της επόμενης θητείας. Αυτό θα πρέπει να το βρουν οι συντονιστές. Μία προσέγγιση για την εξέβρεση συμβιβαστικών λύσεων. Και επαναλαμβάνω ότι δεν είμαι σύμφωνος να στριμώξουμε αυτή την οδηγία μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που μας μένει στη διάθεσή μας. Έκανα πολλές συζητήσεις, έλαβα πολλά σχόλια και πολλές τροπολογίες ε, ε, κατέθεσα προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα επί της αρχής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρόλα αυτά. Γιατί, γιατί από 12 οδηγίες τις συνενώνουμε σε έναν κανονισμό. Εντάξει, να ομαδοποιήσουμε, να συνενώσουμε. Αλλά Μήπως δίνουμε, μήπως αφαιρούμε ε, με τον κανονισμό ένα περιθώριο λιγμών που άρεσε σε πολλά κράτη-μέλη. Μήπως αυτό ε, κρύβεται πίσω από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τα συνενώσει όλα αυτά σε κανονισμό. Αλλά, διρετόρε... Έχω κι εγώ μια ερώτηση για, την, ε, για το διευθυντή Πουγκλέ. Ο κύριος Όσλιγκ το λόγο. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι πρόκειται για συζήτηση. Δεν μπορούμε να βγάλουμε μερικά κομμάτια και να θέσουμε, ε, συζήτηση, να θέσουμε ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρε, αν δεν είναι εδώ πέρα ο εισηγητής, ε, ας μην την κάνουμε τη συζήτηση. Λυπάμαι. Να πω και προς την πλευρά του εισηγητή με επικριτική διάθεση ότι δεν είναι δυνατόν να μην κάνει τη δουλειά του στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να βρούμε με τους ε, συντονιστές μία λύση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Να μην πούμε ότι τελείωσε η συζήτηση. Να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια υπόδειξη για το πώς μπορεί να βελτιώσει την πρόταση που μας υποβάλλει. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί το στόχο μας. Όλα αυτά που κάναμε δεν ήταν συζήτηση για την οδηγία για τους σπόρους. Ο καθένας θα είναι την άποψή του. Αυτό θα πρέπει να το πούμε στους συντονιστές. Θέλουμε να το κοιτάξουμε μέσα στην επόμενη λεωμέλεια, Υπό ποια μορφή να υποδείξουμε μία κατεύθυνση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο λόγο διευθυντή Ποντλέ για να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία τη συζήτηση αυτή. Να ακούσουμε, διευθυντή Ποντλέ. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση παρόλα αυτά. Εάν, επειδή το θέμα είναι πολύ περίπλοκο και είναι πάρα πολλέ οι οδηγίε που ενωπεί ο κανονισμό αυτό εάν δεν μπορέσουμε να διαχωρίσουμε από τα αναπαραγωγικά υλικά του σπόρους και τα καλύψουμε όλα μαζί. Δύο ζητήματα πάνε τελείω διαφορετικά. Τι θα γίνει, κύριε Πουντλέ. Και μετά κλείνουμε γιατί έχουμε και τη συνεδρία των συντονιστών ακριβώ. Κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Είμαι ευτυχής που μπορώ σήμερα να απαντήσω, ακόμη και αν αυτή η συζήτηση δεν είναι επίσημη. Όντως, το θέμα είναι πολύ περιπλοκό και πολύ τεχνικό. Χρειάζεται να έχει κανείς ειδικότατες γνώσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που προκάλεσε τόση συζήτηση το κείμενο αυτό. Να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Μποβέ, του κυρίου Γιάρ, και ίσως να είναι και η δική σας κύριε Πρόεδρε. Γιατί ένας κανονισμός που ασχολείται με 12 οδηγίες. Υπάρχουν δύο απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα 12 οδηγίες ε, ε, καλύπτονται γιατί ακριβώς μιλάμε για οδηγίες που εγκρίθηκαν σε ένα διάστημα 45 ετών. Οι ορισμοί δεν μπορούν να παραμένουν αμετάβλητοι, το ίδιο και οι έννοιες. Οι τεχνικές έχουν αλλάξει, Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των οδηγιών αυτών ως προς τις αρχές τους. Όχι στην προσέγγιση τους ακριβώς. Ε, ακριβώς επειδή είναι οδηγίες, τα κράτη μέλη είχαν μεταφέρει στην εθνική τους νομοθεσία τις οδηγίες αυτές με τρόπο τελείως διαφορετικό πολλές φορές. Ο έλεγχος δεν ήταν αρκετά αυστηρός στο παρελθόν για να δούμε πώς μεταφέρονταν οι οδηγίες στην εθνική νομοθεσία και αυτό οδηγούσε σε σημαντικότατες αποκλήσεις. Αποκλήσεις που δημιουργούν προβλήματα στο ενδοκινοτικό εμπόριο. Μιλάμε για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ε, ελάχιστες, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, που, τον οποίο οι πρόσωποι ήρθαν να μας βρουν και μας ζήτησαν εναρμόνιση. Υπήρχαν πολλά προβλήματα εμπορίας, καμιά φορά και στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, όπου υπήρχαν μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο διαφορετικά από τη μια επαρχία στην άλλη. Μέσα στο ίδιο κράτος, έτσι. Λοιπόν, για αυτούς τους λόγους προτείναμε αυτόν τον κανονισμό που, όπως ξέρετε, ισχύει για όλα τα κάτι μελη υποχρεωτικά, όμως προβλέποντας μια κάποια ευελιξία. Δεν μπορούμε κατά πάντα να τα διευθετήσουμε λεπτομερέστατα σε ένα κανονισμό σαν κι αυτόν. Θελήσαμε μάλιστα στον κανονισμό να συμπεριλάβονται οι διατάξεις που αφορούν τα δάση. Αν και το δάσος έχει τη δική του ζωή. Για όλα τα άλλα φυτά, εκτός των δασικών, μιλάμε για εξουσιοδότηση ποιότητας, ενώ για τα δάση μιλάμε για εξουσιοδότηση προέλευσης του σπόρου βελανιδιάς, του σπόρου οξιάς, του σπόρου ελάτου. Μιλάμε για έλατα του τάδε δάσους της Γερμανίας με τους συγκεκριμένους σπόρους ή την τάδε βελανιδιά από την Ισπανία. Μιλάμε για τι ουσιοδοτήσει τελείω διαφορετικέ, διότι το 80% των ελέγχων είναι πανομοιότυπη, αλλά το 20% είναι ιδιαίτερα ειδική ανάλογα με την προέλευση του δάσου. Για το λόγο αυτό θελήσαμε να συγκεράσουμε τα δάση με τα υπόλοιπα αναπαραγωγικά υλικά. Και επειδή έχω αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να κάνω και μια δική μου αυτοκριτική. Ίσως δεν εκτιμήσαμε αρκετά την ομορφιά αυτού του κειμένου. Επικριθήκαμε σφοδρότατα. Υπόθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να ευνοήσει τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις πολυεθνικές, τις 4-5 πολυεθνικές και να θανατώσει τις ελάχιστες επιχειρήσεις, να θανατώσει τους σπόρους τους, να δολοφονήσει την οργανική και βιολογική γεωργία. Δεν θέλαμε να σκοτώσουμε κανέναν. Δεν θελήσαμε να σκοτώσουμε την εναλλακτική παραγωγή. Όντω, υπάρχει μια σειρά από διατάξει που αφορούν τις ε, λεγόμενες συμβατικέ ε, σπορές, όπου οι νέε ποικιλίε πρέπει να καταγράφονται σωστά. Η αδειοδότηση πρέπει να δίδεται από τις αρχές. Θελήσαμε όμως να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία για τους εμπορευόμενους και να ευνοήσουμε τις νέες ποικιλίε ώστε να μπορούν να καταγράφονται ευκολότερα είτε στους εθνικούς καταλόγους είτε στο κοινωτικό κατάλογο. Προβλέψαμε μέτρα πιο ευέλικτα, πιο ταχαία, πιο εύληπτα για αυτές τις ε, συμβατικές σπορές αλλά και για τις εναλλακτικές, για τις βιολογικές ποικιλίε, τις παραδοσιακέ ποικιλίε, για τις ε, καινοτόμες Προβλέψαμε σαφείς, απλές διατάξεις. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονη κίνηση έπρεπε και οι κανόνες μας να συνάδουν με αυτή την κίνηση. Συμπεριλάβαμε τετερόκλητα υλικά και ετερογενή υλικά. Εδώ Μπορεί κανείς να διευκρινίσει περισσότερο τον ορισμό όπως θέλει η κυρία Κλάς, δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς αυτό. Αλλά θελήσαμε να καταστήσουμε εφικτά όλα αυτά τα συστήματα εμπορίας σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα. Ε, δωρεάν εμπόριο, επιπληρωμή εμπόριο για αυτές τις παραδοσιακές ε, σπορές κατηγορηθήκαμε ότι θελήσαμε να καταστρέψουμε όλα τα καλοπιστικά φυτά, τις παλιές ποικιλίε και αυτό είναι τελείως ψέματα. Συνειδητοποιούμε τι γίνεται, απλώς όσο το εκφράσαμε άσχημα. Το κείμενο αυτό προβλέπει με πολύ σαφέστερο τρόπο ότι τα ισχύοντα τη συνύπαρξη μεταξύ σπορών από συμβατικές ποικιλίε και ήδη οι σπορές για τη βιολογική γεωργία για τις παλιές για τα παλιά είδη, για τα παραδοσιακά είδη, για τις καινοτόμες αγορές. Τέλος, ο κύριος Ταραμπέλα έκανε μια ερώτηση και ζήτησε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα γίνει στην περίπτωση της απόρριψης από την Επιτροπή σας ή από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν διαθεσμικές συμφωνίες, αλλά είναι σαφές ότι το Συμβούλιο έχει προχωρήσει, έχει προχωρήσει στις συζητήσεις του για το κείμενο αυτό. Το Συμβούλιο έχει κάνει προτάσεις βελτίωσης, αλλά δεν σκέφτηκε να απορρίψει τελείως το κείμενο αυτό. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ δυσκολότερο για μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, απέριπταν τελείως το κείμενο. Όμως το Συμβούλιο άρχισε τη δουλειά και ετοιμάζεται να κάνει προτάσεις αλλαγών. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει, αλλά έχουμε την αίσθηση ότι εάν το Κοινοβούλιο στη φάση της πρώτης ανάγνωσης απορρίψει τελείως το κείμενο, το Συμβούλιο θα συνεχίσει τη δουλειά του. Δεν θα αποφασίσω εγώ βέβαια, αλλά Στη δεύτερη ανάγνωση θα έχουμε τα ίδια ζητήματα, με όλες τις δυσκολίες που αυτό μπορεί να επιφέρει στην Επιτροπή σας, την Κομάγκρη και το Κοινοβούλιο. Αυτά είχα να πω, Πρόεδρε, επαναλαμβάνοντας ότι είμαστε απόλυτα πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τα μέλη της Επιτροπής σας για να εξηγούμε, να αποδεικνύουμε την ε, χρησιμότητα του κειμένου αυτού σε σχέση με 12 οδηγίε, να αποδείξουμε ότι δεν θέλουμε να δολοφονήσουμε τι ελάχιστε επιχειρήσει που έχουν λιγότερου από 10 εργαζομένου ή λιγότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ κυκλοεργασιών. Αυτέ είναι το 93% τη αγορά στον τομέα των, ε, της 80% ε, στον τομέα των ε, οποροκυπευτικών, 69% στον τομέα των λαχανικών και 70% στον τομέα των δασών. Άρα υπάρχει ένας τεράστιος ιστός μικρότατων, ελάχιστων επιχειρήσεων που κάνουν τον τομέα αυτό ιδιαίτερα ζωτικό. Ξέρετε ότι η αγορά των σπορών είναι ένας ε, κλάδος με φοβερές εξαγωγές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι φοβερά σημαντικός για το εμπορικό μας ισοζύγιο, διότι 60% των εμπορευόμενων σπορών στον κόσμο προέρχονται από την Ευρώπη. Πρόκειται λοιπόν για ένα τομέα θεμελιώδους σημασία και θέλουμε ακριβώς να διατηρήσουμε για τις μικρότατες αυτές επιχειρήσεις, για αυτές τις μικρομεσαίες ενίοτε τη δυνατότητα να εμπορεύονται είτε σπορές συμβατικές, είτε βιολογικές σπορές για τη βιολογική καλλιέργεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε τον Διευθυντά Πουντλέ και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε όταν συζητήσουμε με τους Σκιώδης και με τους συντονιστές για να δούμε τις απόψεις της Επιτροπής. Και τώρα συνάδελφοι πολύ γρήγορα γιατί μετά δεν θα έχουμε διερμηνείς για τους συντονιστές. Πρέπει να δούμε και το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 120 του κανονισμού σχετικά με την καταπολέμηση της πατάλης στην συνεδρία των συντονιστών να ανακεφαλαιώσω γρήγορα γιατί πρέπει να ψηφίσουμε πολύ σύντομα. Στην ε, συνεδρία των συντονιστών 26 Νοεμβρίου 2013 αποφασίσαμε να ετοιμάσουμε γνωμοδότηση για το θέμα αυτό, για την καταπολέμηση τη επισητιστικής πατάλης. Ε, μια, ένα ψηφίσμα σε μορφή επιστολή που βλέπετε από το άρθρο 120 του κανονισμού. Αυτή η επιστολή πρόκειται να αποσταλεί στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η επιστολή να εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή και να συμπεριλαμβάνει και επιστολή της αρμόδιας ε, επιτροπής της δικής μας δηλαδή, προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Συμπεριλαμβάνοντας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ζητώντα από τον πρόεδρο του ε, Κοινοβουλίου να την παρουσιάσει στην, ε, στο αρμόδιο θεσμικό όργανο. Δηλαδή, ο κύριο Σούλτ να τα πει στον κύριο Μπαρόζο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η γραμματεία τη Άγκρη ετοίμασε ένα σχέδιο τη επιστολή βασιζόμενη στην πρόταση ψηφίσματο που μα είχε απασχολήσει, λαμβάνοντα υπόψη τις προτάσει τη συνεδρίαση των συντονιστών. Σα ζητώ λοιπόν τώρα να μου πείτε αν συμφωνείτε. Την έχετε δει την επιστολή. Συμφωνείτε. Πρέπει να ψηφίσουμε εάν συμφωνούμε και να αποστείλουμε την επιστολή αυτή στον πρόεδρο Σούλτ, ο οποίο θα την ιδιοποιηθεί για να την προωθήσει στον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν αντιρρήσει. Συμφωνείτε όλοι. Πρέπει να ψηφίσουμε όμω. ε. Σας παρακαλώ. Οι παρόντες και οι παρούσες, σηκώστε τα χέρια σα τουλάχιστον. Υψώστε τα χέρια σας. Συμφωνείτε. Διαφωνείτε. Μόνο οι φιλελεύθεροι συνήθω. Α, και ο κύριο ε, Ανιώ. Ευχαριστούμε. Η Επιτροπή σταματά τη συνεδρίασή της. Όχι, όχι, μισό λεπτό, το θέμα άγγινιο είχε ζητήσει να συζητήσουμε κάτι στα διάφορα ο κύριος Άγνιου. Παρακαλώ, Άγνιου. Ευχαριστώ πολύ στα διάφορα. Οι βουλευτέ θα είδαν ίσω ότι έχω διανύμει ένα σημείωμα και έναν χάρτη στην Κομισιόν, την οποία θέλω να προκαλέσω να μας δείξει πώς ένας αγρότης μπορεί πώς να το πω, να συμμορφωθεί με τους πολύπλοκους κανόνες ε, για τα EFAs. Waiting. Για τις επιτρεπόμενες καλλιέργειες έχουμε κάποιους συντελεστές. Μπορεί να δει κανείς που είναι, αυτή είναι αυτά τα EFA, αυτές οι περιοχές και να καταλάβουν πόσο πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει αν αυτοί δεν μπορούν να, τις, τις κομισιόν δεν μπορούν να καταφέρουν να, να υποβάλουν σωστά ζητήσει, πόσο μάλλον ένας Βρετανός αγρότης και που θα χάσει και τις επιδοτήσεις του. Ευχαριστούμε κύριε Άγγινιου. Λάβαμε το σημείωμα. Ε, ε, λίγη συνεδρίαση της Επιτροπής, δύο λεπτά διάλειμμα και παρακαλώ τους να μείνουν.